Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο σημείο της μερικής διάταξης σήμερα είναι να καλωσορίσουμε τον αντιπρόεδρο της Ουγγρικής Κυβέρνησης και Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης Κύριο Τίμπορ Ναβράτσης, τον καλωσορίζουμε, μας τιμά η παρουσία του και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την παρουσίαση του του προγράμματος των δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Κυβέρνησης στον τομέα της δικαιοσύνης για το επόμενο εξάμεινο. Θα τον ακούσουμε 10-12 λεπτά και θα κάνουμε ό,τι κάναμε και χθες. Πρώτος γύρος ερωτήσεων από τους συντονιστές, το πολύ δύο λεπτά ο καθένας πρώτος γύρος απαντήσεων του Υπουργού τι αναφράξεις μετά ανοιχτό δεύτερο γύρο ερωτήσεων από όποιον βουλευτή θέλει να πάρει το λόγο και πάλι θα απαντήσει ο υπουργό. Σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα εδώ για τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας σε σχέση με την δικαστική συνεργασία και ευχαρίστως να σας απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να είμαι λίγο πιο σύντομος από ό,τι μου πρότεινε ο Πρόεδρος, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για ερωταπαντήσεις. Οι στόχοι που έχουμε συμφωνήσει στα πλαίσια της Προεδρίας μας θα ήθελα να τους καταστήσουμε σαφείς, θα ήθελα να επιτύχουμε πρόοδο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. Έτσι όπως το βλέπω εγώ υπάρχουν τρεις τομείς στους οποίους θα θέλαμε να προχωρήσουμε. Καταρχάς, και αυτό είναι ένας από τους γενικού μας στόχου. πρέπει να δούμε την υπηκότητα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε αυτό να φαίνεται, να καταδεικνύεται περισσότερο και σε άλλους τομείς της ε, πολιτικής της Ευρώπης. Έχουμε την ε, Στοκχόλμη και ε, θέλουμε να επιδεχθεί περισσότερο σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα ε, των πολιτών. Η ευρωπαϊκή υπηκότητα είχε πάντα εμπόδια στο δρόμο της και αυτά πρέπει να τα απαλείψουμε. Ξέρω, θα, ξέρω ότι γνωρίζετε ότι ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα και πρόσφατα, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, το, την Παρασκευή στην ε, Ουγγαρία, έγινε μια άτυπη υπουργική συνάντηση και είδαμε την ε, πρόταση της Κομισιόν για την ε, ευρωπαϊκή υπηκότητα και αναφέραμε ποια είναι τα εμπόδια που προκύπτουν από την πρόταση της Κομισιόν. Είδαμε ποια είναι τα βήματα και οι νομικές πράξεις, καθώς επίσης και οι μη νομικές πράξεις, που είναι απαραίτητες για να αρθούν αυτά τα εμπόδια. Επίσης, σε αυτή την άτυπη υπουργική διάσκεψη συζητήσαμε για το πώς θα μπορούμε στο μέλλον πιο αποτελεσματικά να συμπεριλάβουμε και την διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητε του Συμβουλίου και σε όσα κάνει το Συμβούλιο. Παρόλο που η Κομισιόν είναι αυτή που διαπραγματεύεται εδώ και εμείς στο Συμβούλιο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες στοχοθετημένες συζητήσεις. η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έχουμε το θέμα της ε, ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για, την, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε να είμαστε επιτυχείς ως προς αυτό. Βέβαια πρέπει να δημιουργηθούν και κάποιοι εσωτερικοί κανόνες εδώ, εντός της Ένωσης, για να γίνει αυτό, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένα και αυτά βήματα και ελπίζουμε ότι τα βήματα αυτά θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Στον τομέα λοιπόν αυτό μιλούμε για προστασία θυμάτων, για παράδειγμα βοήθεια προς τα θύματα και επίσης ε, πρέπει να, θέλουμε να δημιουργήσουμε και έναν οδικό χάρτη. Θα οργανώσουμε επίσης μία διάσκεψη για την προστασία των θυμάτων και περιμένουμε την ε, ολοκληρωμένο, το ολοκληρωμένο πακέτο της ε, Κομισιόν για τα μέτρα για τα θύματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Επίσης, όταν μιλούμε για ποινικέ διαδικασίες, <coughs> πρέπει να δούμε το δικαίωμα στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση. Υπάρχει μια οδηγία προς αυτό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση, περισσότερη ενημέρωση και περισσότερη ασφάλεια. Επίσης, σε θέματα διαδοχής ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό για να υπάρξει δηλαδή αμοιβαία αναγνώριση των διαφορών συστημάτων διαδοχή. Και επίσης πρέπει να δούμε και γενικώ τι διαδικασίε που υπάρχουν. Πρέπει να απλοποιήσουμε ε, τις διάφορες διαμάχες που προκύπτουν. Ε, υπάρχει η πρόταση Βρυξέλλες 1 που τροποποιεί την, ε, τη δικαιοδοσία στα αστικά θέματα και για να κλείσω κιόλα. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι αρκετά σημαντικό, ίσως να είναι και το πιο σημαντικό. Στενή συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Σίγουρα θα υπάρχουν ε, πολλά θέματα που θα προκύψουν ε, στην διάρκεια των ερωτήσεων και των απαντήσεων, αλλά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούν πολύ καλά, γιατί χωρίς καλή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τίποτα. Εμείς λοιπόν ε, μπορούμε να σας ε, υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε μια ευέλικτη προσέγγιση και επίσης να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη συνεργασία μας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σύντομα και σε ένα καλό αποτέλεσμα όλε αυτέ οι προσπάθειε. Αυτά από μένα και με ευχαρίστω τώρα να ακούσω τι ερωτήσει Σα Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Σα ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομο, και μπορέσατε έτσι να μας συνοψίσετε το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας στον τομέα που εκπροσωπείτε. Οι συντονιστέ τώρα έχουν το λόγο. Ο Σάιμον Μπουσούτου είναι ο πρώτο, εξ του ΕΡΚ. Για δύο λεπτά. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσίαση και για την παρουσίαση του προγράμματός σας. Ε, έχω να αναφέρω διάφορα θέματα. Καταρχήν, ένα που αναφέρατε εσείς, την προστασία των θυμάτων. Από ό,τι κατάλαβα, έχει μπλοκάρει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο πάνω στις ισχυρούσες προτάσεις σε σχέση με την προστασία των θυμάτων που υπευλήθη αρχικά στο Συμβούλιο και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θα προσπαθήσετε να προωθήσετε την πρόταση αυτή εν ώψη σύντομης επίλυσης ή θα περιμένετε την προ... τη νέα πρόταση της Κομισιόν που αναμένεται αργότερα κατά διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας σας. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αθίξω Δεν ξέρω αν είσαστε ο αρμόδιος υπουργό, θα το θέσω εδώ όμως. Πέρσι, αυτή την εποχή, το κοινοβούλιο μας ασχολήθηκε για μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για την ανταλλαγή ε, τραπεζικών στοιχείων, η γνωστή συμφωνία SWIFT. Ένας από τους όρους από τους οποίους εμείς ε, εγκρίναμε αυτή την πρόταση ήταν ότι εμείς θα ότι θα συνεργαζόμαστε για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα δίωξης των τρομοκρατών, ένα EFTP ευρωπαϊκό, ένα θέση προς το αμερικανικό. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ελήφθη αυτή η απόφαση και θα ήθελα να ξέρω τι έχει γίνει. Τέλος, όσον αφορά τις δημοσιονομικές προβλέψεις, θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι ιδέες που θα υποβάλει η Προεδρία εν ώψη της νέες δημοσιονομικές προβλέψεις βέβαια στον τομέα των ε, δημοσίων ελευθεριών και της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος Μωράης. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τα θύματα των ε, εγκλημάτων και για τις δημοσιονομικές προβλέψεις. Από ό,τι κατάλαβα, η Κομισιόν θα υποβάλει σχετικές προτάσεις γρήγορα. Γνωρίζω, Υπουργό, σίγουρα ότι το σώμα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θύματα εγκλημάτων που δεν γνωρίζουν τα διάφορα νομικά συστήματα των χωρών μελών. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιε είναι οι συγκεκριμένε προτάσει που θα υποβάλλετε, ποια δέσμη μέτρων θα υποβάλλετε για τα θύματα των εγκλημάτων. Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση κατόπιν της ακρόασης της περασμένης εβδομάδας στις οποίες υποβάλλατε, ε, απαντήσατε συγγνώμη σε άμεσες ερωτήσεις. Τη ομάδα μου και μου. Πήραμε τώρα μία επιστολή του Επιτρόπου Κρούς που είχε αποστολή στην Ουγγρική κυβέρνηση και που τη γνωρίζετε. Συζητήσει την περασμένη εβδομάδα στην Ακρόαση ζητήσαμε ε, στοιχεία όσον αφορά την ερμηνεία του τι είναι τα ισορροπημένα ΜΜΕ. Μία ανησυχία της Επιτρόπου Κρούς αναφέρει το ότι χρειάζεται ισορροπημένη παρουσίαση από όλα τα ΜΜΕ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η πάποψή σας κατά πόσον αυτό είναι μια, ένας περιορισμός της ελευθερίας πληροφοριών και τι πρόκειται να κάνετε με την επιστολή αυτή της Επιτρόπου. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Άλντε, η κυρία Μπέβερα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που παρουσιάσετε διάφορα θέματα για τα οποία ενδιαφέρεται η Ουγγρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από το θέμα της προστασίας των θυμάτων εθίγει από τους συναδέλφους, δεν θα το αναφέρω, θα περάσω σε άλλα τρία πολύ σύντομα ερωτήματα. Αναφέρετε στο, ε, αναφερθήκατε στο θέμα της υπηκότητας. και ότι εσείς ήδη έχετε σκεφτεί πώς θα πρέπει να ε, ξεπεραστούν τα ισχύοντα εμπόδια. Μπορείτε να αναπτύξετε λιγάκι το θέμα αυτό, να μας πείτε ακριβώς τι έχετε κατά νου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ήταν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα βασικά δικαιώματα μέσα στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου. Και εδώ θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για το όραμά σας σχετικά. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον και πώς η Ουγγρική Προεδρία θα έμπλακει στο θέμα της εποπτείας και πέρα από την εποπτεία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων ΕΕ για το θέμα της συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων. Thank you. For the Greens, Mrs. Argentini. κύριε Σαγκετίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε 6 έως 8 εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι θέμα αυτό της Προεδρίας σας. Μεγάλη τιμή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση κάπως ε, εγκαταλείπεται. Ε, παραδείγματος και στη δική μου χώρα Ανοίγουμε τώρα την συζήτηση για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Κοιτάξτε ας πούμε τι κάνετε εσείς για τα ΜΜΕ που είναι επίσης θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χθε είχαμε τον συνάδελφό σας εδώ και έσυσαμε να συζητάμε το θέμα της καταστολής των διακρίσεων και κατά πόσον αυτό αφορά τα ΜΜΕ και ή όχι κλπ μας είπαν ότι εσείς θα ηγηθείτε ε, τις προσπάθειες αυτής για την υπογραφή της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα ήθελα να ξέρω πώς θα προστατεύσετε τα δικαιώματα αυτά. Κατόπιν, κατόπιν παρατηρήσεων της Ρενάτε Βέμπερ για την προστασία των δεδομένων, ο συνάδελφός σας είπε ότι τώρα ίσως είναι πιο ασφαλές να πάει κανένας από την Ευρώπη στη ΣΥΠΑ παρά να πετάει στο εσωτερικό της Ευρώπης. Και νόμιζω ότι αναφέρεται, το στη, στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για τις πτήσεις. Αν αυτή είναι η ιδέα της Ουγγρικής κυβέρνησης, μπορείτε σας παρακαλώ να αναπτύξετε το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής όταν πρόκειται για θέματα μεταφοράς αεροπορικής. First of all, um, I uh, Με συγχωρείτε, δεν άκουσα δυστυχώ όλα σα τα σχόλια σήμερα το πρωί, γιατί άρχισα να έρθω. Αλλά θα μου επιτρέψετε ίσω να αναφερθώ σε δύο τομεί ε, σύντομα. Ο ένα είναι ε, αυτό το θέμα τη αναλυγή των στοιχείων, ε, ιδίω σε σχέση με το PNR και τι σχετικέ συζητήσει. Όπως ξέρετε, έχουμε μία πρόοδο σε σχέση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζονται τα στοιχεία αυτά. Άρχισε κάπως. Και η Επίτροπος Βάλτστρομ είπε ότι πραγματικά θα υπάρχει ακόμα χρόνος που θα περάσει. Έχουμε όμως πολύ επίγοντα θέματα για το PNR και αναρωτιέμαι κατά πόσον από πλευράς Προεδρίας θα εξετάσουν την ισορροπία αυτή και θα τι θα πρέπει να γίνει ή αν θα αφήσουμε τα πράγματα όσο έχουν. Μετά, όσον αφορά το θέμα των μετακινήσεων ανθρώπων, το αφήνω έτσι πολύ γενικά. Υπάρχουν θέματα σύλλου, υπάρχουν θέματα μετανάστευσης, υπάρχουν θέμα εξωτερικών συνόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το Frontex και τους πόρους που θα χρειαστούμε ίσως για να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να πείτε κύριε Υπουργέ κάποια λόγια για τις απόψεις και προτάσεις σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας πώς θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι τόσοι αντοφατικοί και δύσκολοι τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Γκουε, ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης Ναβάτσης. Εγώ έχω να σας πω ότι είμαι αισιόδοξο για την Ουγγρική Προεδρία. Ότι δηλαδή θα πληρώσει τις προτεραιότητες της, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν πολλές προτεραιότητες. Αναφερθήκατε στα δικαιώματα διαδοχής, στο δίκαιο κληρονομιάς δηλαδή, και στα δικαιώματα των θυμάτων. Αλλά δεν βλέπω τα συγκεκριμένου στόχου που θα πρέπει να επιτευχθούν. Εκτός κάποιες ανακοινώσεις, όχι εναρμόνισης με για τα δικαιώματα αυτά κληρονομιάς. Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις να υποβάλω για τρεις διαφορετικούς τομείς που ανησυχούν πολλούς ε, πολίτες και στη χώρα μου και σε άλλες. Το ένα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπήρξαν κάποιε ειδήσει για τη μερή συμφωνίες με την ΣΥΠΑ ακόμα και μετά που εδόθη η εντολή στην Κομισιόν για να διαπραγματευτεί τη συμφωνία πλαίσιο. Θα ήταν βέβαια πολύ καλύτερο στο Συμβούλιο να υπάρχει μια κοινή θέση που ενδυναμώνει την ευρωπαϊκή δυνατότητα επιβολή των δικών της απόψεων δηλαδή κλπ. Μετά για την ελευθερία έκφρασης, συμφωνώ με πολλές αψαρτήσεις που υποβλήθηκαν και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τις απαντήσεις σας. Αναφερόμαστε στην ελευθερία έκφραση σε όλες τις 27 ε, χώρες, με λίγη μόνο στην Ουγγαρία. Και θα ήθελα να ξέρω, έχετε κάποια ανάλυση να κάνετε για το πώς ε, προχωρά το θέμα αυτό. Γιατί είμαι σίγουρο ότι και το Συμβούλιο θα το εξετάσει το θέμα. Τρίτον, ρωτήσαμε το Συμβούλιο σχετικά με την... Ε, όσο πάει και περισσότερο έντονη ε, ριζοσπαστική τάση στον ε, τομέα της δικαιοσύνης, θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι δικές σας ακριβείς απόψεις, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς τι έχετε κατά νου. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ. Για την EFT δεν βλέπω κανέναν. This group, then we pass... Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στην κυρία Μορβάη για τους μη εγγραμμένους. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εγώ είμαι δικηγόρος, ήμουν δημόσιος κατηγορός και ήθελα να ξέρω για τις απόψεις για τα θύματα, ιδίως τα πιο ευάλωτα θύματα, γυναίκες και παιδιά δηλαδή. Η βία μέσα στις οικογένειες, παραδείγματος χάρη, και εκεί η βία είναι ένα δικό φαινόμενο και πλήττει ακριβώς γυναίκες και παιδιά. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον μέσα στα πλαίσια της προστασίας των θυμάτων θα αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι υπάρχει ενώπιον του Συμβουλίου τώρα μια σύμβαση που προετοιμάζεται για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να στην προσοχή σας. Η Ουγγρική κυβέρνηση δείχνει μια δέσμευση για την προστασία των θυμάτων, αλλά αυτή τη δέσμευση δεν θα λάβει κανένα ε, σοβαρά υπόψη εάν δεν εξεταστούν όλα τα θύματα των εγκλημάτων μεταξύ 2002 και 2010 εγκλήματα που δεν τα γνωρίζει κανένας. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθούμε τι έγινε όταν είπε ο σοσιαλιστική φιλελεύθερη κυβέρνηση η αστυνομία και άλλοι, ακόμα και το δικαστικό σύστημα ε, να το πούμε έτσι, δυσκόλευαν τη ζωή πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, τραυματίστηκαν, απειλήθηκε η ζωή τους από τους τραυματισμούς αυτούς. Είναι σημαντικές αυτές παραβάσεις του, των δασικών δικαιωμάτων και δεν ξέρω αν θα το εξετάσετε το θέμα. Η έκθεση του Γκαγκαϊγκούγιος και άλλων μέσα στα πλαίσια της ε, Ουγγαρίας αυτή τη στιγμή όπου είδαμε ότι οι δικαστές πήραν κάποιες αποφάσεις αντίθεση με οποιοδήποτε δίκαιο. Αυτές ε, δεν έχουν ε, μεταφραστεί σε βασικές γλώσσες όπως ε, αγγλικά ή γαλλικά. Δεν είναι γνωστές λοιπόν αυτές οι, οι περιπτώσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι η εγκουρική κυβέρνηση έχει υποχρέωση και έναντι των δικών της πολιτών και έναντι όλων των πολιτών της Ευρώπης ότι αυτά δεν θα ξαναεπαναληφθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποβολή των ερωτήσεών σας και γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μπω σε λεπτομέρειες όταν μιλάμε για τις προτεραιότητες γιατί νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και διασάφηση των θεμάτων. Θα ήθελα ως υπουργό Δικαιοσύνης να θίξω ορισμένα θέματα, αλλά σε μερικά δεν μπορώ να σας δώσω ίσως ικανοποιητικές απαντήσεις. Ως προς τη, τα εξωτερικά σύνορα και το άσυλο, αυτό είναι θέμα που αφορά το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Πίντερ, του Υπουργού Εσωτερικών. Θα μπορούσα να σας είχε δώσει επαρκείς πληροφορίες. Αν θέλετε όμως, θα μπορούσατε να υποβάλλετε ένα ερώτημα γραπτός έτσι ώστε να σας δώσουμε μια πιο εκτενή απάντηση. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον Υπουργό που ασχολείται με αυτό το θέμα. Εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιό του. Τώρα, ως προς το ερώτημα του κυρίου Ταβάρες. Κύριε Ταβάρες, μιλήσατε για ακραία φαινόμενα, εξτρεμιστικά φαινόμενα και ριζοσπαστικοποίηση γενικότερα. Αυτό δεν αφορά επίσης το χαρτοφυλάκιό μου. Προσπάθησα, θα προσπαθήσω να λάβω απαντήσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Πίντερ, και τώρα για να δούμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις, θα ήθελα να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις που συνδέονται μεταξύ τους για να έχουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ως προς την προστασία των θυμάτων πιστεύουμε ότι πρέπει να κρατήσουμε στάση αναμονής. Δηλαδή να δούμε το πακέτο της Επιτροπής για την προστασία των θυμάτων. Στόχος της Επιτραπής σε αυτό το τομέα είναι να μην δούμε μόνο τους διάφορους ε, νομικούς τομείς, αλλά το πακέτο προστασίας να είναι ένα πακέτο που να υπερκαλύπτει τους άλλους τομείς. Θα θέλαμε όμως να κρατήσουμε στάση αναμονής μέχρι ότου δημοσιοποιηθεί το πακέτο της Επιτροπής. Το δεύτερο προσχέδιο είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν έχει ε, υπάρξει δική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε. Και εάν μιλάμε για την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, το θέμα αυτό θα το κρατήσουμε στην ατζέντα μας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το πακέτο της Επιτροπής. Και Πιστεύω ότι θα επέλθει πρόοδος, διότι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την προστασία των πλέον ευάλωτων κατηγοριών. Πιστεύουμε ότι το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα Μιλάμε για μια ευάλωτη κατηγορία θυμάτων και μαζί με τις γυναίκες θα πρέπει να εντάξουμε και τα παιδιά στην πλέον ευάλωτη κατηγορία. Κατά την ε, προεδρία μας λοιπόν θα θέλαμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Δηλαδή όταν ε, υπάρχει σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη υπάρχει ένα προσχέδιο οδηγίας που πιστεύουμε ότι θα εγκριθεί μέχρι το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας κατά τον Ιούνιο. Τον, ε, κατά τον Ιούνιο, δηλαδή κατά το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ως προς τα δικαιώματα των παιδιών θέλουμε να προστατεύσουμε τις ε, ευάλωτες κατηγορίες και το Μάιο θα υπάρξει μια διεθνής διάσκεψη μέσα στα πλαίσια της ημέρας των παιδιών και θα θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με άλλες μη κυβερνητικές έτσι ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Υπάρχει μια ειδική γραμμή για τα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και υπάρχουν δυστυχώς δύο-τρία κράτη-μέλη που δεν έχουν αυτή την ειδική γραμμή, αυτή τη hotline. Εμείς έχουμε αυτή την ειδική γραμμή για την εξαφάνιση παιδιών και για την αντιμετώπιση του ζητήματος, διότι γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την ευάλωτη αυτή κατηγορία και υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στην Ουγγαρία που προσπαθούν να δώσουν βοήθεια. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Μιλήσαμε για τα στοιχεία επιβατών, για το PNR. Και... Πιστεύουμε ότι θα επέλθει συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε σε σχέση με το σύστημα PNR. Αυτό είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα, διότι θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε το σύστημα PNR. Εδώ μιλάμε για μια ευρύτερη ανάγκη συζητήσεων και διαβουλεύσεων και τα αρχικά βήματα θα γίνουν τον Ιανουάριο στη Βουδαπέστη σε μια διάσκεψη για την προστασία των δεδομένων μέσα στα πλαίσια και άτυπων διαβουλεύσεων έτσι ώστε να συμφωνήσουμε με τις ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας μία βασική τροπή θα δοθεί στην κοινή συνάντηση Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ και πιστεύουμε ότι μπορεί να δοθεί μια νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις αυτές. Γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε ο, ο, ο βασικός διαπραγματευτής αλλά και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα μας βοηθήσουν ως προς την γενικότερη εποπτεία. Από πλευράς Συμβουλίου μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ταχύτερη δυνατή συνεργασία με την Επιτροπή για να σας ενημερώνουμε και για την έκβαση η πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να δούμε τα δικά μας πρότυπα προστασίας δεδομένων για να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με όλα τα δεδομένα. Ο κύριος Μπουζούτιλ μας μίλησε για τις δημοσιονομικές πρόπτικες. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο για να δημιουργήσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών σε σχέση με θέμα με θέματα, με συγχωρείτε, εσωτερικών υποθέσεων. Αυτή είναι και η βασική μας αποστολή με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Άρα θα πρέπει να κινηθούμε πιο κοντά προς τους πολίτες. Και εδώ θα πρέπει να επέλθει ε, συμφωνία και κάποια πρόοδος, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα της ηθαγένειας μας απασχολεί μέσα στα πλαίσια της προώθησης των δικαιωμάτων των πολιτών. Αν δούμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, νομίζω ότι η κυρία Βέμπερ υπέβαλε το ερώτημα σε σχέση ε, από, από πλευράς φιλελευθέρων. Όταν θίξαμε αυτό το πρόβλημα, επήλθε συνένεση για την εξέβρεση μιας λύσης. Αν δείτε τις εσωτερικές δομές του Συμβουλίου, θα πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση τους σε επίπεδο ομάδων εργασίας, σε επίπεδο υπουργών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη φυσικά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχει μια ομάδα που ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και εγώ είμαι επικεφαλής του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Στο μέλλον θα ζητήσουμε από, την Ευρωπαϊκή, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αποφανθεί επί του θέματος. Το Συμβούλιο έχει σαφή πρόθεση να ασχοληθεί με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων με το input που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, Η κυρία Σαρτζεντίνη υπέβαλε ένα ερώτημα το οποίο αν κατανόησα καλά ε, ε, αφορούσε τον ιδιωτικό βίο. Και εδώ η σύμβαση προστασίας δεδομένων που θα συνάψουμε με τη ΣΥΠΑ είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε να μην παραβιάζεται ο ιδιωτικός βίος ή τα προσωπικά δεδομένα. Στο εγγύς μέλλον γνωρίζετε ότι η πρόσβαση στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ύψης της σημασίας, γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα και τον ιδιωτικό βίο. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη την διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ακόμα περισσότερο. Και αυτό το λέω σχετικά με το Συμβούλιο περισσότερο. Όταν μιλάμε όμως για τη συζήτηση μεμονωμένων νομικών πράξεων ή όταν λαμβάνουμε θέση, θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό αφορά και το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Σε σχέση με τον ε, νόμο για τα μέσα ενημέρωσης θα ήθελα να αναφερθώ στην ελευθερία του εκφράζεστε. Ο κύριος Μωράης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Επιτροπή ε, έστειλε μία επιστολή προς την Ουγγαρία σε σχέση με την πλήρη κάλυψη και ίσως διακυβεύεται η ελευθερία του εκφράζεσθε. Όμως υπάρχουν διαφορετικά πολιτισμικά δεδομένα σε κάθε χώρα και οι χώρες λαμβάνουν διαφορετική, έχουν διαφορετική άποψη ανάλογα με τα πολιτισμικά αυτά δεδομένα. Στην Ουγγαρία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν διακυβεύεται η ελευθερία του εκφράζεστε. Αλλά βεβαίως θα λάβουμε υπόψη αυτά που ε, ανέφερε η Επιτροπή και πιστεύω ότι πριν από την εκπνοή της προθεσμίας θα μπορέσουμε να απαντήσουμε επίσημα στα σχόλια της Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε αμφιβολίες γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε την ελευθερία της ελεύθερης έκφρασης. Εάν λοιπόν τίθεται σε κίνδυνο αυτή η ελευθερία θα πρέπει να δούμε το φάσμα των νόμων έτσι ώστε να συμμορφωθούμε με αυτές τις προδιαγραφές γιατί όταν μιλάμε για κάλυψη θα θέλαμε να ληφθούν υπόψη αυτές οι ανησυχίες και να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή κάλυψη γεγονότων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα για αυτό το θέμα της κάλυψης διότι εάν λάβετε υπόψη της, την ομολογία και τις προγενέστερες αποφάσεις δεν υπάρχει παράβαση. Θα πρέπει να υπάρχει εξισορροπημένη ενημέρωση. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να το βλέπουμε ανακανάλι για να δούμε κατά πόσο υπάρχει εξισορροπημένη πληροφόρηση, αλλά να λάβουμε υπόψη μία ευρύτερη εμβέλεια. Δηλαδή δεν μιλάμε για επιμέρους ε, κλιμάκια όπου γίνεται μία επιμέρους μέτρηση αν θέλετε. Θέλουμε μία πιο μία μακρόπνοη θεώρηση του ζητήματος. Αν οι εμπειρογνώμονές μας θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει ευρεία εφαρμογή του νόμου, τότε θα αλλάξουμε το γράμμα του νόμου. Εάν ξέχασα κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Yes, Mrs. Argentini, I beg you Πολύ σύντομα, κυρία Σάρτζεντι. Δεν θεωρώ ότι με ξεχάσατε, αλλά ως προς τις ε, διαπραγματεύσεις με τις ηπα για την προστασία δεδομένων φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις pnr βαίνουν καλώς αλλά ε, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται όμως για ένα πακέτο γιατί μιλάμε για ένα ζήτημα αρχής και αναρωτιέμαι κατά πόσο θα μπορούσατε να μας πείτε πώς μπορούν αυτά τα δύο να παραμείνουν, να ομαδοποιηθούν και να τα αντιμετωπίσουμε μαζί, από κοινού. Δεν θα ήθελα δεύτερο γύρο γιατί έχετε υπερβεί τα δύο λεπτά το χρόνο σας ως συντονίστρια. Δεν θα πρέπει να επεκταθείτε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Αυτό αφορά τον κύριο Ταβάρες το γνωρίζω ότι το θέμα αυτό, δηλαδή ότι μέσα στα πλαίσια των, του χαρτοφυλακίου εσωτερικών υποθέσεων μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και για ε, ριζοσπαστικοποίηση μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε και του συνέρχεστε. Σας ε, ε ευχαριστώ διότι θα ε, ρωτήσετε τον συνάδελφό σας θα υποβάλλεται αυτό το ερώτημα στον κύριο Πίντερ, αλλά το θέμα της ε, ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να μας απασχολήσει, να δούμε δηλαδή κατά πόσο μιλάμε για βία φαινόμενα. Διότι μιλάει για ε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες μπορεί να προσκρούν στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορείτε να μας ε, πείτε κάτι περί αυτού. Ο Υπουργός απαντά. Κυρία Σαρτζεντίνη, εντάχει, θα ήθελα να σας πω ότι οι Αμερικανοί είναι εκείνοι που έχουν καθυστερήσει κάπως μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο με τις ΗΠΑ ε, δεν ε, μπορώ να πω ότι έφταιγε η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, αλλά ούτε και εμείς. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με τους δικούς μας εμπειρογνώμονες και παροτρύναμε την αμερικανική πλευρά να διορίσει έναν εκπρόσωπο με συγκεκριμένη εντολή ως προς το θέμα της ε, προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων. Επίσης, μιλήσαμε για πολιτισμικές διαφορές, άρα εάν μιλάμε για τη λέξη ριζοσπαστικός, αυτό δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία, αφορά και άλλες χώρες. Η λέξη αυτή έχει ένα συγκεκριμένο σημενόμενο και νομίζω ότι ως προς το θέμα φορολόγησης ή άλλους ε, τομείς υπάρχουν διαφοροποίησεις που θα πρέπει να ε, εξεταστούν εκ του σύνεγγυς. Ο ριζοσπαστικός αυτός χαρακτήρας δεν είναι απόλυτα σαφής. Αν μιλάμε τώρα για ακραία φαινόμενα, για ε, εξτρεμισμό και αν το χρησιμοποιούμε ως συνώνυμο του του ριζοσπαστικού αυτού χαρακτήρα, τότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι εννοούμε. Δηλαδή κατά πόσο κανείς δημιουργεί, χρησιμοποιεί τις φιλετικές διακρίσεις οποιοδήποτε άλλο μέσον για να οδηγήσει τη χώρα σε μία δικτατορία. Αν μιλάμε όμως για ριζοσπαστικές ε, αλλαγές, αυτό δεν σημαίνει και εξτρεμιστικά φαινόμενα. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο γύρο και έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό μελών που ζήτησε το λόγο. Θα τους αναφέρω. Infeld, Mrs. Romero Lopez, Mr. Romeva, Mrs. Bauer, Mrs. Angelilli, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano, Mrs. Becerril, Mr. Papa Nicolau and Mr. Foss. So I'll understand that the list is closed. I, I see You also want to be part of this? Yes, Papadopoulou? Papadopoulou? Yes, then I'm going to close it down and I... Κλείνουμε τώρα το κατάλογο και σας παρακαλώ να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να μείνετε στο όριο του ενός λεπτού ο καθένας. Γιατί έχουμε και ψηφοφορίες, έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη, οπότε να δώσουμε το χρόνο στον Υπουργό για να απαντήσει. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την ε, παρουσία του. Διάβασα με προσοχή το πρόγραμμα της ε, Ουγγρικής Προεδρίας και με βάση και την προσωπική σας δραστηριότητα για το μέλλον μιλήσατε για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Βλέπω ότι ως προτεραιότητα έχετε το θέμα των θεωρήσεων με την Ρωσία και Μολδαβία καθώς και Ουκρανία. Δεν μιλήσατε όμως για την αμοιβαιότητα θεωρήσεων ως προς πέντε κράτη-μέλη έναντι των ΗΠΑ και του Καναδά, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να δράσετε άμεσα για να προωθήσετε ε, την αμοιβαιότητα σε σχέση με την Κύπρο, Τσεχία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Δηλαδή να υπάρχει αμοιβαιότητα. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Δύο πράγματα με ικανοποίησαν από αυτά που είπε ο Υπουργό. Καταρχά ότι πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι πρέπει να γίνουν αυτά βήματα υπέρ των πολιτών. Αντί λοιπόν να έχουμε ένα γραφειοκρατικό ρολόι που χτυπά στα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τι νομικέ τα νομικά εργαλεία έτσι ώστε να να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δομές. Πρέπει να εφαρμοστεί και η οδηγία για την διακριτική μεταχείριση. Τώρα, ο, αυτός ο αντικρουόμενος α, νόμος που έχετε για τα ΜΜΕ, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι τα ΜΜΕ θα πρέπει να ε, ε, σέβονται την ε, αξία του γάμου και της οικογένειας και μετά υπάρχει ένας ορισμός, ένας νέος ορισμός το, του γάμου και, του, και της οικογένειας ε, στο σύντομα που το περιορίζει σε άντρα και γυναίκα. Και μάλιστα όταν, όταν παρουσιάστηκαν εικόνε δύο ε, γκέι αντρών στην τηλεόραση, αυτό θεωρήθηκε ότι καταπατά το Σύνταγμα και τον ορισμό της οικογένειας του γάμου κτλ. Θα ήθελα να μου πει ο Υπουργό. Ε, η, η Ουγγρική Προεδρία τι ακριβώς θα κάνει ώστε να γίνουν πραγματικότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και για, τους, ε, για την κοινότητα των ομοφιλοφίλων στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό τη. Η κυρία Ρομέρο. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα θέμα ταμπού στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το αντιμετωπίζετε. Μιλάμε για βία κατά γυναικών και παιδιών. Έχουμε πολύ υψηλούς αριθμούς. Μπορείτε να μας πείτε ποιες γυναίκες, ποιος είναι ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί βία στη χώρα σας Εάν θέλετε να μπορέσει να δράσει το παρατηρητήριο, θα πρέπει να ξέρουμε τα αριθμητικά στοιχεία της Ευρώπης, διότι μιλάμε για 2.500 γυναίκες στην Ισπανία, αλλά δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το ένταλμα προστασίας. Γνωρίζω τις δηλώσεις της Επιτροπής και γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα αφορά και ασφαλιστικά μέτρα, αλλά η Επιτροπή δεν έχει θίξει το θέμα των ασφαλιστικών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι υπάρχουν 100.000 ε, εντολές προστασίας και έχουμε πολλές γυναίκες από την Ουγγαρία θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα κατά γυναικών από την Ουγγαρία, υπέρ συγγνώμη γυναικών από την Ουγγαρία και αν επιστρέψουν στην Ουγγαρία θα τύχουν τις ίδιες προστασίες. Ε, Κύριε Υπουργέ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Να επαναλάβω ένα ερώτημα που ήδη τέθηκε για την ε, μη διακριτική μεταχείριση και τη σχετική οδηγία. Ε, το παρακολουθούμε και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων προεδριών και με την Ισπανία και με το Βέλγιο το είδαμε. Στη δική σας την, στη δική την Προεδρία πόσο ψηλά στις προτεραιότητες σας είναι το θέμα αυτό. Γιατί μιλήσατε και για την ηθαγένεια και είπατε ότι αυτή είναι η προτεραιότητά σας και μιλήσατε και για τους Ρωμά αλλά και αυτή η οδηγία έχει σχέση με του Ρωμά. Οπότε, ω προ αυτό, θα ήθελα να μου πείτε πώ ακριβώ προτίθεστε να προχωρήσετε στην εκπόνηση ε, αυτή τη οδηγία, στην ε, ε, διεκπαιρέωσή τη, γιατί ξέρουμε ότι κάποια κρατημέλη ακόμη ανησυχούν. Πώ θα διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση, θα υπάρξει κάποιο χρονοδιάγραμμα για να την να διαχειριστείτε και μπορούμε να περιμένουμε μέσα αυτό το εξάμεινο να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα ω προ αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Δύο ερωτήματα έχω να θέσω στον Υπουργό. Στην τελευταία ολομέλεια μιλήσαμε για την διεθνή διαδοχή. Διορθώνει η μιλήτρια για, τη διεθνή, για τις διεθνείς υιοθεσίες και υπάρχει ένα πλαίσιο για τις ε, ε, υιοθεσίε και μιλούμε για την α, ε, αναγνώριση, μη αναγνώριση μεταξύ κρατών μελών. το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης εμπορικών και αστικών υποθέσεων επίσης είναι αυτό που αναφέρατε πιο πριν. Θα συμπεριλάβετε και τις υιοθεσίε σε αυτό. Και δεύτερον, η ηθαγένεια. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια καταρχάς. Προφανώς ε, εφαρμόζεται εδώ η επικουρικότητα, γιατί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια ε, συνδέεται και με την ηθαγένεια κράτους μέλους. Σε κάποια κράτη-μέλη ε, αυτή η δυνατότητα υπάρχει, αυτή η πρακτική, αλλά κάποιος χάνει την ηθαγένειά του σε κάποια κράτη-μέλη εάν ζητήσει ηθαγένεια από άλλο κράτος μέλος. Τώρα, αν μιλούμε για τρίτες χώρες, είπα ας πούμε και τα λοιπά. Ας πούμε αν υπάρχει ένας ε, πολίτης ε, Αμερικανός, αν θέλει να γίνει Ευρωπαίος θα χάσει την Αμερικανική ειδικότητα και θα, ε, έχει μόνο την ε, Ευρωπαϊκή. Αν θέλετε λοιπόν πείτε μου πώς ακριβώς προτίθεστε να το δείτε το θέμα αυτό. Και επίσης, στην περίπτωση των ευρωπαϊκών κρατών, Πώς μπορούν δύο κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα σύστημα που ε, διπλό, διπλής ηθαγένειας που όμως η μία ηθαγένεια αναιρεί την ύπαρξη της άλλης. Ε, ναι, σας παρακαλώ να μείνετε στα όρια τα χρονικά γιατί έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα για να μπορέσει και ο υπουργό να απαντήσει. Η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό διότι υπογράμμισε ότι η οδηγία για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των παιδιών και κατά της πορνογραφίας είναι μία από τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας. Και εγώ στο τέλος αυτής της συνεδρίασης θα έρθω σε επαφή με έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου για να ορίσουμε αυτό το πλαίσιο που αφορά τον τριμερή διάλογο. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να υποβάλω σε σχέση με, αυτά που είπε η κυρία Μπάουερ καταρχήν, κατά πόσον θα υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων για τα παιδιά προσιοθεσία. Διότι όπως μας είπε η κυρία Μπάουερ, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα που ορίζει, το, οριοθετεί το θέμα των εγκαταλειμμένων παιδιών και τα οποία θα μπορούν να υιοθετούνται από τις ε, χώρες, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά βεβαίως από την αναγνώριση των εγγράφων και τις δικαστικές αποφάσεις. Μία άλλη ερώτηση αφορά το εξή Θα υπάρξει μία ενημέρωση και αναθεώρηση σε σχέση με την εθνική νομοθεσία και ως προς την απαγωγή παιδιών από έναν γονέα στους μικτούς γάμους, διότι πολλές φορές απομακρύνονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά. Thank you, Mr. President. Mr. Vice Prime Minister, welcome. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε. Η οριζόντια οδηγία για την μη διακριτική μεταχείριση είναι σαφώ, όπω είπαμε και οι πολύ σημαντική για μα. Έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει μια θέση και το Συμβούλιο δεν κινείται. Είπατε ότι σα ενδιαφέρει. Συμφωνείτε να πούμε ότι ας πούμε σε δύο μήνες θα επανέλθετε εδώ στην Επιτροπή μας και θα μας δώσετε μια αναφορά για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις στο ζήτημα αυτό. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, πέρα από τις καλές προθέσεις πρέπει να έχουμε και κάτι απτό στα χέρια μας από το Συμβούλιο. Οπότε θα με χαροποιήσω πάρα πολύ αν συμφωνούσατε να επανέλθετε σε δύο μήνες και να μας πείτε τι γίνεται. Επίσης, οι φυλακές και οι συνθήκες κράτησης. Η Διεθνής ε, Σύμβαση για την Ανθρώπινη Μεταχείριση και την, απα... και την ε, ε, μη, και, την, και, τα, και μη ύπαρξη βασανιστήριων ε, λέει ότι θα πρέπει να, γίνονται, να υπάρχουν επισκεπτήρια και ότι θα πρέπει να ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων. η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική βεβαίως μέσα στα κράτη-μέλη και οι συνθήκες σε πολλέ είναι, σε πολλές χώρε είναι πραγματικά τραγικές. Η Κομισιόν έχει μία πράσινη βίβλο γι' αυτό. Έχετε πρόθεση εσείς να το συζητήσετε αυτό στο Συμβούλιο με του υπόλοιπου συναδέλφου σα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλφάνου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αποβάλω το εξή ερώτημα. Ξέρετε ότι οι μη κυβερνητικέ και οι κοινοί γνώμοι ανησυχούν για την Προεδρία σας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ως προς τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, όπου υπάρχει και ένας νόμος που απαγορεύει τον γάμο μεταξύ ομοφιλοφίλων. Θα ήθελα να μου δώσετε πληροφορίες και για μια άλλη ιδιάζουσα κατάσταση. Αφορά την πρόεδρο του Media Council και θα ήθελα και πληροφορίες ως προς τις αρμοδιότητες της Προέδρου γιατί διάβασα πληροφορίες όπου λέγεται ότι η πρόοδος ακολουθεί ομοφοβική στάση. Έχει απαγορεύσει ορισμένες ε, εκπομπές και ε, μου φαίνεται κάπως περίεργη η θέση της. Έχει απαγορεύσει και την κυκλοφορία ορισμένων περιοδικών. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Θα ήθελα ως από κοινού συντάκτρια με την κυρία Ρομέρο να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας Θυμάτων. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τη θέση σας εγώ ως μέλος της ε, Επιτροπής ε, Γυναικών. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα προστασίας των θυμάτων και ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών. Μιλήσατε επίσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Με χαροποιεί αυτό, αλλά θα ήθελα να μου πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά πόσο θα υποστηρίξει και τα θύματα τρομοκρατικών πράξεων γιατί ζητούν απονομή δικαιοσύνης και τίποτα περισσότερο. Παπα Ο κύριος Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Ε, θα αναφερθώ σε ένα πιο ειδικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία. Το προηγούμενο διάστημα εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη, αναφέρω ενδεικτικά την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, ε, ύποπτα δέματα δέματα που υπήρχε υπόνοια ότι περιείχαν εκρηκτικές ουσίες. Και ε, τα δέματα αυτά είχαν διάφορους παραλήπτες, μέχρι και την καγκελάριο της Γερμανίας, αρχηγούς κρατών, πολλές πρεσβείες και ε, μας απασχόλησε και μας απασχολεί έντονα το ζήτημα αυτό. Και το ερώτημα είναι, σκοπεύει το επόμενο διάστημα η Ουγγρική Προεδρία να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Θεωρεί πως το πρόγραμμα της Επιτροπής για την πρόληψη και την προετοιμασία και τη διαχείριση των, ε, ε, συνεπειών στον τομέα της τρομοκρατίας μέχρι το, 2013 επαρκεί. Θα κάνουμε ενδεχομένως κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά το ρόλο της Europol. Ευχαριστώ πολύ. Hello. Yes. Uh, you have overemphasized the strengthening. Ενισχύσατε, είπατε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και ότι αυτό θα είναι μία από τις ε, προτεραιότητές σας. Θα εξετάσετε το καθεστώς των ε, ε, των καταφυγίων και το πώς κρατούνται εκεί οι γυναίκες, ε, πώς, ε, επίσης ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι συνθήκες που κρατούνται οι γυναίκες και τα παιδιά σε τέτοια καταφύγια. Επίσης η παιδική πορνογραφία, υπάρχει περίπτωση να δούμε καλές πρακτικές από τη μία ε, και την άλλη, ή κάποια άλλη χώρα. Επίσης ελευθερίες και δικαιώματα των πολιτών τονίσατε ότι όλοι οι πολίτε τη Ευρώπη θα πρέπει να έχουν την, τουλάχιστον τη βασική προστασία των δικαιωμάτων του. Το δικαίωμα τη ελευθερία που ακόμη το αρνούνται σε κάποια κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όμω τι γίνεται. Ο κύριο Φω, ευχαριστώ. Μετά από τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι, δύο σύντομα δικά μου. Καταρχά υπάρχουν κάποιες σκέψεις ε, για τα ενάρξη των δεδομένων, για τη συλλογή δεδομένων ε, για τους ε, επιβάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης το, το ένταλμα έρευνας. Τι γίνεται με το θέμα αυτό, θέλετε να το προωθήσετε, το έχετε βάλει στην, στις σα. ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη ποικιλία και μεγάλο αριθμό ερωτήσεων. Ε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κάνει έτσι μια σύνοψη ο, ο υπουργό για να μπορέσει να απαντήσει σε όλους και έπρεπε να έχουμε ήδη από τις 10 ξεκινήσει τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι σχετικά σύντομο και ο υπουργό για να μπορέσουμε όλοι να ικανοποιηθούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα βάλω τα δυνατά μου. Δεν ε, θέλω να απαντήσω σε, μια, σε ερωτήσεις μία προς μία. Θα απαντήσω έτσι ομαδικά. Ε, μιλήσατε για την γενική οδηγία, την οριζόντια οδηγία για την μη διακριτική μεταχείριση. Αν ε, μιλάμε για το Ουγγρικό Σύνταγμα, το Σύνταγμα απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση επί τη βάση ε, πολιτικών, πεπιθήσεων, ε, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ. Τώρα, αν μιλούμε για την γενική οριζόντια οδηγία, αυτή μπαίνει στα πλαίσια στις του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ η Ουγγρική Προεδρία θέλει να προχωρήσει, αλλά δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες ω προς αυτό, γιατί αυτό είναι σε άλλου Συμβουλίου Ορμοδιότητα, οπότε δεν μπορώ εγώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτού. Επίσης, άλλη μια, ε, συζήτηση που, άλλη μια ερώτηση που τέθηκε ήταν οι υιοθεσίες. και αν γίνεται να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων που λαμβάνονται για τις αεροθεσίες. Εάν δείτε την διάσκεψη της Χάγης, μιλάει για τη σύμβαση περί υιοθεσιών, που νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Οπότε, νομίζω ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα. Τώρα, αν μιλούμε για βία εντό τη οικογένεια, ενδοοικογενειακή βία εναντίον των γυναικών ή παιδιών, συνθήκε ε, στις ε, κράτησης στις ε, φυλακές. Γενικώ, το όλο θέμα της προστασίας των θυμάτων θα θέλαμε λίγο να το περιμένουμε. Θα θέλαμε να δούμε τι θα βάλει η Κομισιόν στο τραπέζι, τι θα προτείνει. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις πληροφορίες που θα έχουμε, τους κανόνες. Θέλουμε να έχουμε καταρχάς μια πλήρη εικόνα για την προστασία των θυμάτων και θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τέτοιες ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες. Τέθη ένα ερώτημα για τις φυλακές και τις συνθήκες και το κατά πόσο ο Ευρωπαίος Δημοσιολογητής μπορεί να δει τι γίνεται στην καταστήση στις περιπτώσεις αυτές. Πρόσφατα ο ε, Ούγγρος διαμεσολαβητής έκανε μία έρευνα για τις ε, φυλακές στην Ουγγαρία, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ο εθνικός συνήγορος του πολίτη να μελετήσει το τι γίνεται στις ε, ε, φυλακές στο κάθε κράτος μέλος. Επίσης, ετέθη ένα ερώτημα για τις θεωρήσεις και την αμοιβαιότητα. Στη Βουδαπέστη, την Παρασκευή, θα συζητηθεί από τους εμπειρογνώμονες. Ε, θα υπάρξουν λοιπόν επιδρογνώμονες οι οποίοι θα δούνε ακριβώ αυτό το θέμα τη αμοιβαιότητα και των θεωρήσεων. Μετά, το ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Εντολή για την Προστασία. Ε, πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο δεν έχει ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για το θέμα αυτό. Οπότε δεν έχουμε την απαιτούμενη υποστήριξη. Βεβαίως, ε, εμείς ως Προεδρία θα πρέπει να κάνουμε τον διαμεσολαβητή, τον διαιτητή λίγο μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορώ να σας δώσω εκτίμηση για το τι θέλουμε, τι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά ίσως η Κομισιόν στα μέσα της Προεδρία μας να μπορεί να υποβάλει ένα πλήρες πακέτο για την προστασία των θυμάτων Η κυρία Μπάουερ ρώτησε για την ηθαγένεια και το ποια είναι η δική μου γνώμη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει το δικαστήριο. Πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο εάν ε, υπάρχουν τέτοια θέματα ερμηνεία σε ό,τι αφορά τους ε, νόμους περί ηθαγένεια στα κράτη-μέλη. Η κυρία Αλφάνο. Νομίζω ότι έχει καλύτερη πληροφόρηση από μένα για τις δραστηριότητε ε, του Προέδρου του Συμβουλίου για τα ΜΜΕ. Γιατί ούτω ή άλλω και εκεί υπάρχουν, ε, και στον τομέα αυτό υπάρχουν δικαστικέ αποφάσει. Εντάξει, πάντα μπορεί κανεί να προσβάλλει τι αποφάσει αυτέ ε, στο δικαστήριο, τι αποφάσει που παίρνει το σχετικό συμβούλιο. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ να έχει γίνει κάποια τέτοια αναφορά για, για άσχημα σχόλια ή για κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως αυτά δεν ξεφεύγουν από τα ΜΜΕ. Στην, ΣΥΠΑ υπήρχε μια σχεδόν ναζιστική οργάνωση που διέδιδε το μίσος και μιλούσε συχνά εναντίον των Εβραίων και προωθούσε τέτοια αισθήματα μίσους αλλά αν προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, ειδικά στα πλαίσια του, των ΜΜΕ, ένας από τους στόχου του νόμου για τα ΜΜΕ είναι αυτός ακριβώ. ότι πρέπει όντως να, σταματήσει, ε, να σταματήσουν τέτοιου είδους ε, εκφράσει. Τώρα να απαντήσω στο θέμα, για το θέμα της θερμοκρατίας. Δεν είναι μόνο το θέμα της θερμοκρατίας, είναι και το θέμα της προστασίας των α, θυμάτων. Ε, συμφωνώ λοιπόν με αυτό που λέτε. Είναι καλό που οι κυβερνήσεις έχουν διάφορα, διάφορους υπουργούς που ασχολούνται για το θέμα αυτό, ώστε να μπορούν όλοι συγκροτημένα να αντιμετωπίσουν το θέμα. Επίσης πρέπει να τονίσουμε το ότι είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα θύματα ώστε να υπάρχει μια πιο ισόρροπη κατάσταση σε όλο το φάσμα των κυβερνήσεων. Αυτά για το θέμα αυτό. Κυρία Παπαδοπούλου, αυτό ε, που λέτε συνδέεται και με την προστασία των δεδομένων. Οπότε μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν ως προς αυτό. Για την βία κατά των γυναικών, κατά των παιδιών. Ε, θα πρέπει να περιμένουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν. Τώρα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που αν τα θεμελιώδη δικαιώματα παραβιάζονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ε, οι πολίτες μπορούν να πάνε στο δικαστήριο. Υπάρχουν επίσης πολλά διεθνή φόρα στα οποία μπορεί κανείς να ε, απευθυνθεί πριν ξεκινήσει ε, να χρησιμοποιεί τα ένδικα μέσα. Ο κύριος Φως επίσης μίλησε για την ανταλλαγή PNR. Δεν έχω κάποια α, πληροφόρηση ως προς αυτό. Δεν ξέρω να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Αν ε, έχετε λίγη υπομονή, μπορώ να το ψάξω και να σας απαντήσω γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρομέρα, έχετε υπόψη ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο όμω. Σα παρακαλώ να είστε σύντομοι κατά δυνατόν. Δεν μου δόθηκε απάντηση από τον Υπουργό. Ποιος είναι ο αριθμός θυμάτων στη χώρα σας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία. Θα ήθελα να σας πω ότι το ευρωένταλμα Μάλλον το έγγραφο της Επιτροπής δεν μιλά για αναγνώριση ασφαλιστικών μέτρων. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσετε, να ταχθείτε υπέρ της ευρωεντολής και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εξέτασα άλλα πράγματα ε, τη σεξουαλική βία κατά των παιδιών ε, αλλά δεν έχω στοιχεία αριθμητικά όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών. Θα ζητήσουμε από μη κυβερνικέ οργανώσεις και οργανώσεις προστασίας των γυναικών να μας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για να σας ικανοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, λέει ο Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις αυτές και για την πρόθεσή σας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. θα παρακολουθήσει στενά την Προεδρία. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Dear colleagues, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας. If you want to take your seats, please. So that we can proceed because... Καθίστε σας παρακαλώ για να συνεχίσουμε. Γιατί έχουμε αρκετή καθυστέρηση. Please. We're having now a number... Λοιπόν, έχουμε μία σειρά ψηφοφοριών τώρα. Πέντε στο σύνολο. Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Θα τις πάρουμε τη μία μετά την άλλη. First one is included in the order of the day as point 12. Λοιπόν, το πρώτο σημείο ψηφοφορίας είναι το σημείο 12. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Σύνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λίχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013. Λοιπόν, έγκριση σχεδίου σύστασης. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Άρχεται ηλεκτρονικά. No, not working. Now it's working. Okay, the vote is open. No, no, no, it's not. Άρχεται η ψηφοφορία. Not working. Not working. We're going to see how many. Για να δούμε. Πόσοι ψήφισαν. Τώρα λειτουργεί το σύστημα. Ωραία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 49. 43 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Όχι. Ωραία. Δεύτερη ψηφοφορία τότε. Δεύτερο θέμα. Σημείο 13. Προσχώρηση του Λίχτενστάιν στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ελβετίας σχετικά με τη σύνδεση Ελβετίας στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σέγγεν. Έχουμε πάλι την έγκριση ενός σχεδίου σύστασης μπροστά μας. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε της ψηφοφορίας. Στα νέα ψηφίσαντες, 48 υπέρ, κανένας κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. having a third vote. Voting the Τρίτη ψηφοφορία, σήμα 14. Προσχώρηση Λίχτενστάιν, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ελβετία σχετικά με το προσδιορισμό κράτου που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτηση ασύλου που υποβάλλεται σε κράτο μέλο ή την Ελβετία. Έχουμε πάλι μια έγκριση σχεδίου σύσταση. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. Σαράντα δύο υπέρ, τέσσερις κατά και τρεις αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο σύστασης. Πολύ ωραία. Now, I guess we're moving Point number 15. Τώρα περνάμε στο σημείο 15. Point number 15 relates the agreement που αφορά τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχίας διαμονής για τους κατόχους κοινών διαβατηρίων. Ψηφίζουμε. Now the vote is closed. Πέραση ψηφοφορία. 44 υπέρ. 2 κατά. 3 αποχέ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Και. Πέραση ψηφοφορία. Με 16. Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Βραζιλία για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση βραχία διαμονή για του κατόχου διπλωματικών, υπηρεσιακών ή επισήμων διαβατηρίων. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 3 απαχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα... Now we're moving. Και τώρα, περνάμε. Now we're moving. If you please, to the Λοιπόν, περνάμε στο σημείο που ανεβλήθη χθε το πρωί. Διαδικασία ενία αίτηση για άδεια παραμονή και εργασία. Αυτό έχει αναπαυθεί στην Επιτροπή μας βάσει του άρθρου 563 ε, του κανονισμού του σώματος που λέει ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα επαναπέμπεται, η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει την ακολουθητέα διαδικασία και προφορικά ή γραπτά θα το παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μέσα σε μια περίοδο που αποφασίζεται από το Κοινοβούλιο και που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο μήνες. Στην περασμένη συνεδρία στις 10 Ιανουαρίου Πρόεδρο ζήτησα από την Γραμματεία να ελέγξει από τις υπηρεσίες της Ανομέλειας τι θα πρέπει να κάνουμε για να επιστρέψουμε στο, στην Ολομέλεια με μια πρόταση που λαμβάνει υπόψη το αίτημα της Επιτροπής Εργασίας Απασχόλησης να παραμείνει συνδεδεμένη μαζί μας για το θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, η κυρία Ματιού, η συγγήτρια Λίμπε, θα μας εξηγήσει κατά πόσον η ακολουθητέα διαδικασία που προτείνει θα πρέπει να συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή. Μετά τη συζήτηση θα ψηφίσουμε για να ορίσουμε την θέση της Επιτροπής για τη διαδικασία. Κυρία Ματιέ, θέλετε να μας εξηγήσετε την άποψή σας. Α, διαδικαστικό. Ή μετά την κυρία Ματιέ. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο τη Επιτροπή Απασχόληση, την κυρία Μπερέ. Η κυρία Ματιού έχει το λόγο. Ah, Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Κατώ ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου για την έκθεσή μου για την ενιαία αίτηση, είχε αποφασιστεί να επαναπευθεί το θέμα στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 3 του κανονισμού. Μετά από διαβούλευση με τι ε, υπηρεσίε, ε, νομοθετικού συνονισμού και τι υπηρεσίε Ολομέλεια, ιδίω τον κύριο Ντόνσταν, μας ελέγχθη το εξή για τη διαδικασία. Το άρθρο 56.3 λέει ξεκάθαρα ω σε περίπτωση της επαναπομπή Επιτροπή η αρμόδια Επιτροπή αποφασίζει τη διαδικασία που θέλει να ακολουθήσει και το παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο γραπτά ή προφορικά μέσα στη προθεσμία που ορίζει αυτό που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ λοιπόν, που είναι η αρμόδια Επιτροπή, πρέπει να εκφραστεί πάνω στην ακολουθητή διαδικασία. Όσον αφορά το περιεχόμενο του κειμένου, η Επιτροπή Απασχόληση θα πρέπει να εμπλακεί σε όλα τα σημεία του κειμένου που είναι δική της αρμοδιότητας και που πρέπει να τροποποιηθούν για να επιτευχθεί πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, Προτείνω διαδικαστικά να υποβληθεί στην Επιτροπή μας αρχές ε, Φεβρουαρίου ιδανικά μια συμβαστική πρόταση που θα βασίζεται στην ψηφοφορία της Ολομέλειας όπου θα τροπηθούν κάποια σημεία για να επιτευχθεί πλειοψηφία. Και προτείνω να τροποποιηθεί ένα τμήμα το που θα είναι το μόνο που θα ψηφιστεί και το υπόλοιπο ο μπλοκ να ψηφιστεί στην Ολομέλεια για τα σημεία που δεν ήταν δηλαδή αντικείμενα τροποποίησεων. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις αυτές, από τις διαβουλεύσεις μου με τις πολιτικές ομάδες υπάρχουν μόνο λίγα σημεία αποκλειστική αρμοδιότητα τη Επιτροπή ΛΥΒΕ πρέπει να τροποποιηθούν για να επιτευχθεί πλειοψηφία. Εν κατακλείδη, η Επιτροπή Απασχόληση δεν χρειάζεται να παρέμβει στην προετοιμασία του συμβαστικού κειμένου. Γιατί οι τροπολογίε τη δική αρμοδιότητα που ψηφίστηκαν στην δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν. Τέλο, προτείνω να υποβληθεί σήμερα σε ψηφοφορία αυτή η ε, διαδικασία που προτείνω. Εάν εγκριθεί η διαδικασία αυτή, θα έλεγα ότι η συζήτηση για τα σημεία που ήταν αντικείμενο διαφωνίας στην Ολομέλεια να ξεκινήσει αμέσως, να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας αρχές Φεβρουαρίου και να υποβληθεί η συμβαστική πρόταση στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Before we hear from the chair Τώρα θα ακούσουμε την ε, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης για να γνωρίζουμε σε ποια τμήματα της πρωτοβουλίας θα διαχωρίσετε το περιεχόμενο για να ξέρουμε ποια τμήματα θα ψηφίσουμε, ως προς τη διαδικασία δηλαδή. Πρόκειται για τα άρθρα που αφορούν το επιπρόστατο έγγραφα και τα, τους πίνακες αντιστοίχησης. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί με καλέσατε από πλευράς τη Επιτροπής μου για το κοινό αυτό θέμα που μας απασχολεί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όπως ξέρετε, έχουμε συντάξει μια επιστολή προς τον πρόεδρο Λένε για κατανομή αρμοδιοτήτων των δύο επιτροπών μας στις 8 Μαρτίου 2010 για καταμερισμό ή επιμερισμό αρμοδιοτήτων και έγινε λόγος για το 9, 12, 15 και 16 αιτιολογικές σκέψεις 2 β 3β, 12 εκτός από την πρώτη παράγραφο και παράγραφο 13. Αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν όταν εξετάσουμε τις ψηφοφορίες επί της εκθέσεως Ματιέ στις 12 Δεκεμβρίου. Βλέπω ότι αυτή η πρόταση απερίφθη κατά την τελική ψηφοφορία Είχαμε 306 ψήφους υπέρ, 350 κατά και 25 αποχές. Απορρίφθηκε η έκθεση Ματιέ επειδή με βάση τις τροπολογίες του ΕΛΚ φτάναμε στην αρχική θέση του Συμβουλίου μέσω τροπολογιών. 30 λοιπόν τροπολογίες εγκρίθηκαν επί της εκθέσεως Ματιέ. επί των 30 ε, τροπολογιών που εγκρίθηκαν και οδήγησαν στην απόρριψη της πρότασης, οι 15 σχετίζονταν με το τμήμα που σας προανέφερα, δηλαδή που αφορά τη βάση τη συμφωνία μας, όπου είχαμε και την υποστήριξη του κυρίου Λένε. Οι 15 τροπολογίες αφορούν αποκλειστικά την έκθεση Αλεσάνδρο Φέρκας και αφορούν σημεία επί της ουσίας, δηλαδή τα άρθρα 2, 3, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αφενός και αφετέρου το άρθρο 12 που αφορά τις εξαιρέσεις κάλυψης όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα για υπηκόους τρίτων χωρών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι θέμα δική σας ευθύνης ή αν υπάρχει διχογνωμία ως προς την ερμηνεία, το θέμα θα αφορά την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, συνταγματικών, με συγχωρείτε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι αμφισβητήθηκε κατά την τελική ψηφοφορία. Άρα δεν μπορούν να ανοίξουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις γιατί επί της ουσίας θα πρέπει να δείτε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΛΥΜΠΕ. Η κυρία Ματιέ, χωρίς να ε, μας πει συγκεκριμένα ποια άρθρα θα ξανα ε, συζητηθούν, μιλά περισσότερο για τους πίνακες αντιστήχησης και για ορισμένα άρθρα. Άρα νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για να δείτε κατά πόσο μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια ως προς θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας η Επιτροπή επί που αποφαίνεται επί της ουσίας δεν αναγνωρίζει τα θέματα της Επιτροπής, της Συνδεδεμένης Επιτροπής. Στις 3 ε, και 18 Ιανουαρίου σας έστειλα μία επιστολή αναφέροντας ότι η Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να ασχοληθεί με τα θέματα δικής της αρμοδιότητας και τα οποία άλλαξαν άρδιν μετά τις τροπολογίες του ΕΛΚ οι οποίες εγκρίθηκαν όσον αφορά το στάδιο διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Ως προς την ερμηνεία του άρθρου 56.3 νομίζω ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτό το άρθρο χωρίς να το συσχετίσουμε με, τα άρθρα 50, με το άρθρο 50 που ακριβώς αναφέρει ότι η διαδικασία της Επιτροπής, της Συνδεδεμένης Επιτροπής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία του, της έκθεσης αυτής και νομίζω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα πρέπει να αποφανθεί σε σχέση με τις δύο συνδεδεμένες επιτροπές και την επιμέρους αρμοδιότητά τους. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο κατά τη συζήτησή μας να δώσουμε το λόγο και στην εισηγήτρια, στον εισηγητή έτσι ώστε να αποφανθεί. Προτείνω να ακούσουμε τους συντονιστές και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδεις. D'accord. Ευχαριστώ, λέει ο εισηγητής, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω επί του θέματος, το οποίο είναι ύψης της σημασίας. Αφορά όχι μόνο αυτή την Επιτροπή, αλλά και άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό νομίζω ότι στην απόφαση που θα σας ε, προταθεί από την κυρία Ματιά θα πρέπει εσείς να αποφασίσετε για ένα θέμα που αφορά και άλλες επιτροπές. Γιατί μιλάμε για δικαιώματα πολιτών που ποτέ δεν συζητήθηκαν από αυτή την Επιτροπή. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, διότι στην πρόταση που άκουσα αναφέρεται ότι η Επιτροπή Απασχόλησης είναι συνδεδεμένη Επιτροπή, αλλά ε, παρερμηνεύοντας το γράμμα του κανονισμού αποκλείεται αυτή η Επιτροπή έμπρακτα. Γι' αυτό υπάρχει αποκλισμός μια συνδεδεμένης Επιτροπής. Εγώ μιλώ εξ όλων των συντονιστών της Επιτροπής Απασχόλησης γιατί για λόγους προηγουμένου δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Εάν ήταν αντίστροφη η κατάσταση, δηλαδή εάν εγώ έπρεπε να αποφανθώ επί της ουσίας και η ΛΥΜΠΕ ήταν συνδεδεμένη επιτροπή, ποτέ δεν θα μπορούσα να θεωρήσω ότι θα λύσω τα θέματα της άλλης επιτροπής ψηφίζοντας τη δική μου επιτροπή. Είναι θέμα μεγάλης ευθύνης, διότι πρόκειται για θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν σε αυτή την Επιτροπή. Πρόκειται για μια διαδικασία που οδηγεί σε μια διένεξη μεταξύ των δύο Επιτροπών, διότι εάν θέλουμε να σώσουμε μία πλειοψηφία από τις, ε, από τις συντηρητικές ομάδες, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να χαλάσουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο επιτροπών. Το να γίνει αναπομπή στην ε, Ολομέλεια θα ήταν λάθος. Μην ψηφίσετε κάτι που αφορά την Επιτροπή Απασχόλησης, διότι αύριο μπορείτε να βρεθείτε στην αντίστροφη θέση και δεν θα, αρέσει, δεν θα σας άρεσε κάτι τέτοιο να αντιστραφούν οι όροι. Εγώ έχω μεγάλη θητεία κοινοβουλευτική και στη χώρα μου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε η πλειοψηφία να μην κατατροπώσει την μειοψηφία. Μπορεί να αλλάξει τον κανονισμό, αλλά δεν μπορεί να γίνει ψηφοφορία για την ερμηνεία ενός κανονισμού. Αυτό το κάνουν οι πρόεδροι των επιτροπών ή οι νομικές υπηρεσίες των κοινοβουλίων. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Μιλάμε για διαδικασίες, για διαδικαστικά θέματα τα οποία αφορούν νόμους που δεν την χάνουν ερμηνείας. Νομίζω ότι σήμερα έχετε βεβαίως την δύναμη, αλλά δεν, έχετε, δεν θα έχετε δίκιο αν προχωρήσετε και ερμηνεύσετε έτσι τον κανονισμό. Ας ακούσουμε τώρα το, τους συντονιστές. Uh, θα μιλήσω εξ ονόματος της ε, ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά θα αναφερθώ σε ένα ευρύτερο ζήτημα. Το πρώτο θέμα είναι ότι η δυνάμη του άρθρου 56.3 εμείς είμαστε η Επιτροπή Αναπομπής Δηλαδή παραπέμπεται το θέμα εκ νέου σε εμά. Και αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. αυτό το άρθρο είναι σωστό, το 56.3. Όταν όμως μιλάμε για νομοθετήματα και μιλάμε για θέματα μετανάστευσης, νόμιμης μετανάστευσης, όπου η Επιτροπή Απασχόλησης είναι συνδεδεμένη Επιτροπή, και τα θέματα αυτά συζητήθηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης και ψηφίστηκαν και όταν ψηφίζονται από την Ολομέλεια θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το θέμα αφορά και, τις ε, άλλες, ε, και τα άλλα θέματα ως προς εποχικούς εργαζόμενους, το, ε, την ενιαία άδεια παραμονής και ούτω καθεξής. Εάν το άρθρο 50 δεν ακολουθηθεί κατά την πρώτη ανάγνωση, τότε είναι ε, επίπλαστη η κατάσταση και θα πρέπει η Επιτροπή Απασχόλησης να είναι εκ νέου συνδεδεμένη και να μπορεί να υποβάλει τροπολογίες. Και θα ήθελα οι άλλες πολιτικές ομάδες να μην κοιτάξουν μόνο την τρέχουσα πολιτική της ε, μεμονωμένης άδειας, αλλά να δούμε ολόκληρο το πακέτο της νόμης μετανάστευσης δυνάμει του άρθρου 54. Οι σκιώδεις ήρθαν σε αυτή την επιτροπή και κατέβαλαν μία προσπάθεια να κατανοήσουμε εμείς ότι το άρθρο 50 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Η νομική επιτροπή εκφράστηκε παρομοίως, όπως είπαν και οι συντονιστές. Άρα δεν μιλώ ως πολιτική ομάδα, μιλώ ως επιτροπή. Έχει σημασία πώς θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή Απασχόλησης Δυνάμει του άρθρου 50. Και αν θέλετε αυτό να το διαχωρίσετε από θέματα συνεργασίας θα ήταν λάθος Θα πρέπει να τηρήσουμε αυτό τον κανόνα, να αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία για να αποσαφωνιστεί νομικά το θέμα του άρθρου 50. Θα έπρεπε να είχε γίνει κάτι τέτοιο κατά την πρώτη ανάγνωση και να ήταν συνδεδεμένη η Επιτροπή Απασχόλησης. Θα ήθελα αυτό να αποσαφινιστεί. Προτείνω αναστολή της πληροφορίας μέχρι ότου αποφανθεί η νομική επιτροπή και να το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Mrs. Weber. Thank you very much, Chair. I'd like to, uh... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να θυμίσω στην Επιτροπή ότι αυτή δεν είναι η πρώτη συζήτηση που κάνουμε για το φάκελο αυτό μετά την απόρριψή του από την Ολομέλεια. Και πρέπει να το πω αυτό, γιατί δεν θέλω οι συνάδελφοι που δεν ήταν εδώ στην πρώτη συζήτηση που κάναμε στην Επιτροπή μας να θεωρήσουν ότι εμείς ε, δρούμε ως ασυνείδητοι. Ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Τότε αποφασίστηκε ότι θα προσπαθούσαμε να έχουμε νομική γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία. Λάβαμε τη νομική γνωμοδότηση λοιπόν της νομικής υπηρεσίας και η γνωμοδότηση ήταν σαφής. Πρέπει να προχωρήσουμε σύμφωνα με αυτά που θα μας πει ο εισηγητής. Η διαδικασία αυτή υποβάλλεται σε ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Οι συζητήσεις λοιπόν για το αν πρέπει να συνδέσουμε αυτή την ε, πρόταση μετά την ε, απόρριψή της στην ε, Ολομέλεια ήταν ήδη, έχει ήδη γίνει στην Επιτροπή μας. Έχουμε τη συνεργασία βάσει του άρθρου 50, αλλά μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πτυχών ε, ασκολί ε, ένας, ε, μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμός στοιχείων έγινε αντικείμενο ζήτηση από την Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτά όμως που είναι, μπορούν να είναι συζητήσιμα, μπορούν να τύχουν επεξεργασία και μπορούν να ψηφιστούν, μπορούν να, ε, πρέπει να έρθουν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το δει εδώ η Επιτροπή μας το φάκελο αυτό. Αυτή είναι η δική μου έτσι, εντύπωση για τα όσα έχουν ε, υποθεί μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σέβομαι απόλυτα την Επιτροπή Απασχόλησης και όσους την εκπροσωπούν εδώ σήμερα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι εδώ υπάρχουν δύο σαφή θέματα που πρέπει να παραμείνουν σαφή και ξεχωριστά. Το ένα είναι το θέμα της διαδικασίας το δεύτερο είναι το ουσιαστικό της υπόθεσης. Και θα ήθελα να πω κάτι και για τα δύο. Γιατί νομίζω ότι θα είναι λάθος να τα μπερδεύσουμε αυτά τα δύο. Για τα διαδικαστικά. Στη ζωή κάποιος πρέπει να αποφασίσει. Και οι διαδικαστικοί κανόνες, ειδικά η παράγραφος 56, άρθρο 56 διορθώνει ο εισηγητής, ε, παράγραφος 3 λέει σαφώς ποια είναι η Επιτροπή καθήλυν αρμόδια να αποφασίσει για τη διαδικασία. Και στο άρθρο αυτό λέει σαφώς ότι είναι η αρμόδια Επιτροπή που θα πρέπει να ε, αποφασίσει και για τη διαδικασία. Οπότε δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένα, καμιά, καμιά σύγκρουση ε, επιτροπών είναι οι κανόνε που δείχνουν ποια επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για τα διαδικαστικά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα θέμα ερμηνεία. Δεν πάμε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων όταν ένα ε, άρθρο είναι απόλυτα σαφές και μας λέει απλά και ξεκάθαρα ότι η Επιτροπή, η αρμόδια, η, ε, η υπεύθυνη Επιτροπή είναι η αρμόδια Επιτροπή και ξέρουμε όλοι ότι η αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ανεξάρτητα από το τι λέει το 50. Οπότε, επί της διαδικασίας τα πράγματα είναι σαφή. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι η αρμόδια Επιτροπή. Οπότε, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Επί της ουσίας τώρα. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια η γνωμοδότηση και δεν έτυχε τη στήριξη τη πλειοψηφία. Μπορεί ο καθένα να δώσει διαφορετική ε, ερμηνεία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όμω φαίνεται ότι είναι σαφέ ότι ο λόγο για τον οποίο καταψηφίστηκε η έκθεση ήταν το θέμα των επιπλέον εγγράφων, που είναι ένα ζήτημα το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ. Οπότε, ακόμη και επί της ουσίας, και πάλι είναι σαφές ότι το θέμα είναι θέμα της ΛΥΜΠΕ. Χωρίς εδώ να θέλω να πω ότι ε, αρνούμαστε να αναγνωρίσουμε τις ε, αρμοδιότητες της ε, Επιτροπής Απασχόλησης στα υπόλοιπα άρθρα. Φυσικά τις έχει και γίνονται σεβαστές, αλλά δεν αποφασίζουμε επί της ουσίας σήμερα. Αποφασίζουμε επί της διαδικασίας. Και για τη διαδικασία η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι αυτή που είναι αρμόδια. Κλείνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλω να πω ότι όταν κάτι είναι σαφές, δεν ζητούμε ερμηνεία. Γιατί θα καταλήξουμε να, το σαφές να το κάνουμε ασαφές. Αυτό που χρειάζεται είναι να προχωρήσουμε γιατί πλησιάζει επικίνδυνα η προθεσμία και ένα τέτοιο πακέτο όπως αυτό όπου ακόμη μπορούμε να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση είναι σημαντική. Ε, είναι σημαντικό και πρέπει το συντομότερο δυνατόν να το λύσουμε. Ευχαριστώ. Uh, Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Σάιμον και η κυρία Βέμπερ. Είναι απόλυτα σαφές ότι η θέση είναι αυτή που αναφέρουν. Το άρθρο 56 είναι σαφές, αλλά το 56 δεν είναι απλώς ένα άρθρο που μας βοηθάει είναι ένα άρθρο που υπάρχει για να μας ε, καθοδηγεί στο πώς θα προχωρήσουμε. Οπότε, αν δεν ακολουθήσουμε το άρθρο 56, στην περίπτωση αυτή, τότε νομίζω ότι θα έχουμε και σε μελλοντικέ περιπτώσεις παρόμοιε ε, δυσκολίες λόγω σύγχυση Η Επιτροπή απασχόληση. είχε την ευκαιρία τη, τους δώσαμε την ευκαιρία να, κάνει, να κάνουν τη συζήτησή του. και τα σημεία πίεση. Ε, για τα οποία ε, αναπέμφθη ε, η έκθεση αυτή είναι σημεία τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ. Οπότε εμείς θα αποποιούμασταν τον ευθυνό μας εάν δεν κάναμε όπως προτείνει ο Σάιμον και το υποστήριξε και η κυρία Βέμπερ. Εγώ υποστηρίζω πλήρως την άποψη αυτή και ως Επιτροπή νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη υπευθυνότητα και να ε, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια άλλη πολιτική ομάδα θέλει να πει κάτι που δεν, αν δεν έχει εκφραστεί ακόμα η κυρία Έρμστ. Äh, Βλέχτηκα λίγο και είχα ζητήσει από την αρχή το λόγο, Πρόεδρε. Λοιπόν, διαπιστώνω ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές θέσεις στην αίθουσα και ερμηνείες του κανονισμού. Η Επιτροπή Απασχόλησης και οι δύο εκπρόσωποι της κατέστησαν σαφές ότι και στην Επιτροπή Απασχόλησης υπήρξαν ε, διαφορετικές ερμηνείες για τον κανονισμό, για το συγκεκριμένο άρθρο. Τώρα, αν ισχύει αυτό, για ένα τέτοιο σημαντικό φάκελο, που μπορεί να οδηγήσει και σε προηγούμενο, ε, είναι απαραίτητο να έχουμε σαφήνεια σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για το πώ θα το διαχειριστούμε. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα και εμένα με μπερδεύει πολύ. Υπάρχουν πολύ διάφορες πολιτικές θέσεις. Εγώ δεν θέλω να αποφασίσουμε σήμερα. Αλλά σήμερα ας ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος από το να πάμε στην νομική υπηρεσία, να πάμε να την ακούσουμε την νομική υπηρεσία, να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δεν πειράζει να περάσει μια εβδομάδα, αλλά θέλουμε να έχουμε νομική σαφήνεια γιατί θα χρειαστεί και σε μελλοντικέ περιπτώσει να προχωρήσουμε όπω σήμερα. Οπότε δεν θέλουμε σήμερα να ψηφίσουμε, να συμφωνήσουμε για την, για την πρόταση αυτή. Δεύτερον, έχω τεράστιο πρόβλημα με το ποιε είναι οι βασικές προτάσεις ε, τροπολογίες της κυρίας Ματιέ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Θέλουμε να τι εξετάσουμε αυτέ τι μεμονωμένε προτάσει. Και για να τι εξετάσουμε θέλουμε στην ομάδα μα χρόνο. Και σίγουρα παρόμοιο χρόνο θα χρειαστούν και οι υπόλοιπε ομάδε να δουν ποιε είναι οι βάσει αυτέ που έχετε στην πρότασή σα. Τρίτον, δεν γίνεται η Επιτροπή ε, ε, Απασχόληση να μείνει απ' έξω. Δεν το θέλουμε καθόλου αυτό γιατί θα ήταν τεράστιο λάθος και για μελλοντικές αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σε μια παρόμοια περίπτωση στην ε, Ολομέλεια, όπως έγινε και τώρα. Υπήρξαν πολύ σημαντικές τροπολογίες, βαρύνουσες τροπολογίες και υπάρχουν και μέσω του ε, κανονισμού ε, σύνδεσμοι με την Επιτροπή Απασχόληση. Η Επιτροπή Απασχόληση πρέπει οπωσδήποτε να ε, συμπεριλαμβάνεται στην όλη αυτή τη διαδικασία. Η πρότασή μας λοιπόν είναι σαφής. Να αναβάλουμε την απόφαση, να ακούσουμε την νομική υπηρεσία και βάσει τα όσα μας πει η νομική υπηρεσία να αποφασίσουμε. Uh, Ο Ταβάρες. Σύντομα. Ακούσαμε πολύ σημαντικά νομικά επιχειρήματα από την κυρία Μπερές. Ακούσαμε και θέματα που αφορούν την κοινοβουλευτική συνεργασία από τον κύριο Σέρκας, που επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί προφανώ θα βρεθούμε και στο μέλλον σε παρόμοια περίπτωση. Είναι κρίμα που η ψηφοφορία στην Ολομέλεια ερμηνεύεται με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι η κυρία Ματιέ θεωρεί ότι ψηφίσαμε κάτι μόνο και μόνο για να ε, θέσουμε, για να καταστήσουμε σαφή τη θέση της Λίβη, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και θα ήθελα να απαντήσω απευθείας σε κάτι που είπε ο Σάιμον. Είπε ότι αν κάτι είναι σαφές, πρέπει να το ακολουθήσουμε. Ναι, αλλά αν κάτι είναι τόσο σαφές στους κανόνες, δηλαδή αν η ΛΥΜΠΕ είναι σαφές το τι πρέπει να κάνει, δεν χρειάζεται να μας, να μας ανησυχεί αν θα εμπλακεί κάποια άλλη ε, ε, επιτροπή, γιατί και η άλλη επιτροπή, σύμφωνα με αυτούς τους ξεκάθαρους κανόνες, υπέρ μας το ψηφίσει. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία από αυτού. Το κοίταξα με τους ε, ε, συμβούλους μας, το κοιτάξαμε τους συμβούλους μας και δεν βρήκαμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε μελετήσει λοιπόν την ε, γνωμοδότηση αυτή. Αν υπάρχει, νομίζω ότι θα πρέπει να την, να τη δούμε. αν δεν υπάρχει, να τη λάβουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία, Πρόεδρε. For the Greens, Madame Okay, thank you, President. Um, I must... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήμουν η Σκιώδη στην Επιτροπή, αλλά και συντονίστρια στην Επιτροπή ε, Απασχόληση για το θέμα αυτό. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα ακούστηκαν. Πρέπει όντως να το δούμε πολύ προσεκτικά γιατί μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο. Έχουν υπάρξει και άλλες εκθέσεις μέσα σε αυτό το πακέτο για διάφορες άλλες πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής, πολλές από τις οποίες μάλλον συνδέονται με τα δικαιώματα εργασία και με τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία επίση είναι καθολική, καθολική αρμοδιότητα τη Επιτροπή Απασχόληση. Ένα από αυτά, ένα, από, ένα στοιχείο που θα μπορούσε να μα ωφελήσει μέσα στην συζήτηση αυτή των δύο επιτροπών είναι να γίνει περισσότερη συζήτηση μέσα σε αυτέ τι δύο επιτροπέ αντί να ε, τα πούνε μόνοι τους, η μόνη της, η καθεμιά επιτροπή στα, στο εσωτερικό της. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα θέματα που θα, που θα αποφασιστούν εδώ για το πεδίο εφαρμογής θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις και στις απόψεις των, όσων, των μελών της Επιτροπής Απασχόλησης για την ενιαία άδεια συγκεκριμένα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Και η θέση της ομάδας μου είναι να επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα και να αποφασίσουμε τότε. Εφόσον θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε πώς συνδέεται ο κανόνας 50 με τον κανόνα 56 και όχι μόνο ο 56, ίσως να καταλήξουμε στην ίδια θέση με τον εισηγητή, που προτείνει, με αυτή που προτείνει ο Σάιμον. Αλλά, ε, εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει έτσι μια ανησυχία για, την, για τον καθορισμό προηγούμενου τώρα, το οποίο μπορεί μετά να μας παγιδεύσει στο μέλλον, ε, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Now, there's some, some point over there. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να προχωρήσουμε ε, με βάση τον τονισμό. Το, αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι μιλούμε για πραγματικές καταστάσεις. Το είπε και ο, η Βέμπερ και ο Σάιμον και ο συνάδελφος Κέρκοπ. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Εγώ ζητώ να ψηφίσουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καμία άλλη συζήτηση. Ο κύριος Θέρκας, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εντάχει ως Επιτροπή και για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μπουζούτιλ μίλησε για την βασική επιχειρηματολογία. Το 56.3 όμως δεν μιλά για την Επιτροπή επί του μιλά για την αρμόδια Επιτροπή. Άρα η όλη επιχειρηματολογία είναι για κάτι που οι άλλοι δεν γνωρίζουν. Θα ήθελα να διαβάσετε το 56.3. Δεν μιλά για επιτροπή επί της ουσίας. Μιλά για την αρμόδια επιτροπή. Έχουμε να κάνουμε με δύο αρμόδιες ε, επιτροπές, διότι το άρθρο 56 αναφέρεται στις αρμόδιες επιτροπές. Άρα δεν αληθεύει αυτό που είπε ο κύριος Μπουζούτιλ για τον κανονισμό. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπο να ακούσουμε τις διαφορετικές ε, απόψεις, διότι υπάρχει διχογνωμία για ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες από νομικής ε, άποψης, αν διαβάσουμε το 56.3 και το 50 του κανονισμού. Νομίζω ότι ακούσαμε εκείνους που θεωρούν ότι η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει για τον κανονισμό και ακούσαμε και ισχυρισμούς που υπενθυμίζουν ότι το θέμα της αρμοδιότητας ε, αφορά την Επιτροπή επί της ουσίας για την ενιαία αίτηση και είναι ένα θέμα που αφορά την Επιτροπή Λίμπε και Αμπλουά. Και αυτό αφορά το τρίτο κεφάλαιο, τα άρθρα του τρίτου κεφαλαίου. Άρα δεν μιλάμε μόνο για το προηγούμενο που θα δημιουργηθεί, εάν δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια από πλευρά συνδυασμένη εφαρμογής αυτών των δύο άρθρων. Υπάρχουν διαφορετικές οδοί για να διασαφηνίσουμε αυτό το σημείο έγινε λόγος για την Νομική Επιτροπή και για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για να διασαφηνίσει αυτό το ζήτημα της συνδυασμένης ερμηνείας. Υπάρχουν συντονιστές που ζήτησαν να γίνει τώρα ψηφοφορία και συντονιστές που ζήτησαν την αναβολή. Προτείνω λοιπόν ε, προτείνω να ψηφίσουμε, εάν θέλουμε να ψηφίσουμε την πρόταση της κυρίας Ματιέ ή να αναβάλουμε για μία εβδομάδα την ψηφοφορία, κάτι που θα μας επέτρεπε να διασαφηνίσουμε αυτό το θέμα από νομικής πλευράς και να ζητήσουμε κατά πόσο είναι σκόπιμο να ξανανοίξει η συζήτηση επί των άρθρων της Επιτροπή, του κεφαλαίου 3. Θα ψηφίσουμε τώρα για το αν θέλουμε τώρα να γίνει ψηφοφορία ή να αναβάλουμε για μία εβδομάδα. Για να δούμε τι θέλει η Επιτροπή ε, επί της πρότασης Ματιέ. Ψηφίζουμε τώρα αν τασόμαστε υπέρ του να ψηφίσουμε τώρα ή να αναβάλουμε την ψηφοφορία για μία εβδομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω από την ανάταση χειρών θα ψηφίσετε ναι αυτοί που θέλετε να ψηφίσουμε τώρα και θα ψηφίσετε όχι όσοι πιστεύετε ότι πρέπει να αναβάλουμε για μία εβδομάδα την ψηφοφορία μέχρι ότου να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Ναι, όσοι θέλετε να ψηφίσουμε τώρα λοιπόν. Όχι όσοι θέλετε να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Αρχίζει η ψηφοφορία. I don't have a voting card. Δεν έχω κάρτα, λέει ο ομιλητής, να με συμπεριλάβετε όμως. Now the vote is closed. No. No. The vote is still open. Χρειαζόσαστε περισσότερο χρόνο για να ψηφίσετε. Πέρας. 27. 27 υπέρ, 20 κατά, άρα θα ψηφίσουμε ως προς την ακολουθητέα διαδικασία. Εντάξει κυρία Ματιέ. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα απαντώντας την πληθώρα παρεμβάσεων. Από τη μία πλευρά μεταξύ 10 Ιανουαρίου και σήμερα, όπως υπενθύμησε η κυρία Βέμπερ, έγιναν συνεδριάσεις σκιωδών που οργάνωσα εγώ. Διαπραγματευτήκαμε το όλο θέμα. Μίλησαμε και με τον Αλεχάνδρο Θέρκας και με άλλους συναδέλφους. Θα ήθελα να πω ότι ήρθαμε σε επαφή με τις υπηρεσίες ε, νομικού συντονισμού και θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα ήθελα να θίξω τα άρθρα για την απασχόληση διότι υπάρχει πλειοψηφία στην ομάδα μου. Δηλαδή τα άρθρα που αφορούν την Επιτροπή Απασχόλησης, λέει η ομιλήτρια και διακόπτη, τα άρθρα που αφορούν την Επιτροπή της Απασχόλησης δεν θα θυγούν. Παρακαλώ μην μιλάτε εκτός μικροφώνου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η Ολομέλεια αποφάνθηκε σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής σαφώς. Δεν αποφάνθηκε μόνο η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η Ολομέλεια αποφάνθηκε για όλες τις τροπολογίες. Ακόμα και αν στην τελική ψηφοφορία ήταν σαφές ε, η έκβαση. Μπας περιπτώσει έχει αποφανθεί το σώμα, κατά σαφέστατο τρόπο. Άρα τώρα θα γίνει η ψηφοφορία. Όπως πρότεινε η κυρία Ματιέ. Κατά πόσον δηλαδή θα ακολουθήσουμε την διαδικαστική ερμηνεία που μας εξήγησε η κυρία Μάτιε με την κοινή ερμηνεία των άρθρων 50 και 56.3. Δεύτερη ψηφοφορία για τη δική της πρόταση. Ποιοι συμφωνείτε, όσοι συμφωνείτε ναι, όσοι διαφωνείτε θα ψηφίσετε όχι. Now Πέρας. Again. Πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. 27 υπέρ, 20 κατά. Άρα εγκρίθηκε η πρόταση της εισηγήτριας κυρίας Ματιό. colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Point the order of the έχουμε ακόμα άλλα δύο σημεία στη μέση διάταξη. Σε μία ώρα. Παρακαλώ να λοιπόν, συνεργαστείτε. Really? So it's an hour. Even less than that. We got half an hour to go. Λοιπόν, μισή ώρα έχουμε και δύο σημεία. Παρακαλώ συνεργαστείτε λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 17. Τροχοποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχείριση Περιθυντική Συνεργασία στο εξωτερικό Σύνολο των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινό Frontex. εισηγητής ο συνάδελφο Σάιμον Μπουσούτιλ. Πρέπει να συζητήσουμε τις τροπολογίε που έχουν υποβληθεί για το Frontex. Η προθεσμία υποβολής ήταν 14 Δεκεμβρίου. 185 τροπολογίε υπήρχαν μόνο. Πήραμε και την τελική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Λουάκη ΑΦΕΤ που υιοθετήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, μετά θα ακούσουμε την Επιτροπή και την Προεδρία για τις πρώτες αντιδράσεις και θα έχουμε και τη δυνατότητα συζήτησης. Κύριε Μπουζουτήλ, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομα στην εισαγωγή μου. Η εργασία στην Επιτροπή ΛΥΜΕ είναι πολύ πιο εύκολη όταν τα περισσότερα μέλη φύγουν από την αίθουσα. You have my sympathy. Ε, σας κατανοώ βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Εγώ υπέβαλα 68 στην αρχική μου πρόταση έκθεσης και 186 περαιτέρω υπευρέθησαν, δηλαδή σύνολο 254 τροπολογίες. Αρχίζω τώρα να λυπούμε που ενθάρρυνω του αδέλφους να υποβάλουν τροπολογίες, αλλά τι να κάνουμε. Πραγματικά πρέπει να τους ευχαριστήσω για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουν σε αυτό το φάκελο. Είχα ήδη μια σειρά συναντήσεων με σκιώδεις ηγητές και σκοπεύω να έχω και άλλες, γιατί ελπίζω ειλικρινά ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ε, ισχυρό, ενοποιημένο κείμενο που θα παρουσιάζει την θέση όλων των κομμάτων για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Γενικά θα ήθελα να σας ε, τι μορφή είναι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Σύντομα μόνο και μετά θα περιμένω να ακούσω τις αντιδράσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου και φυσικά και να ακούσω τις ερωτήσεις των συναδέλφων. οι περισσότερες τροπολογίες ασχολούν τα βασικά δικαιώματα, όπως το περιμέναμε. Αυτές τις τροπολογίες μπορώ να τις υποδιαιρέσω σε τρεις τύπους. Μια πρώτη προσέγγιση, αν θέλετε, που ακολουθείται από εμέ και το ΕΛΚ και την ομάδα ΕΛ, ΑΛΤΕ, μια προσέγγιση που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία αρχική δήλωση που θα αναφέρει ρητά ότι τα βασικά δικαιώματα θα πρέπει να διχάνουν σεβασμού από την υπηρεσία αυτή πάντα. Και να σταματήσουμε εκεί. Αυτή είναι η μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση θέλει να εισακάγει μία αναφορά στα ε, βασικά δικαιώματα σε κάθε άνθρωπο του κανονισμού περίπου. Αυτή είναι η δεύτερη προσέγγιση που ακολουθεί η γκου και η πράσινη. Υπάρχει μια τρίτη προσέγγιση που είναι στο μέσο θα έλεγα που ακολουθούν οι σοσιαλιστές. Βάσει αυτού θέλω να πω ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τροπολογία για τα βασικά δικαιώματα της ΑΛΤΕ που προτείνει να υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή που θα διαβουλεύεται πάση στιγμή με την Frontex και θα συμπεριλαμβάνει τις αρμόδιες οργανώσεις του τομέα. Ταυτόχρονα, μου αρέσουν και κάποιες από τις συμπληρωματικές αναφορές στα βασικά δικαιώματα σε επιμέρους άρθρα που έχουν υποβάλει οι σοσιαλιστές. Ελπίζω λοιπόν να θα μπορέσουμε πραγματικά να βρούμε λογικό συμβιβασμό για το θέμα αυτό ούτω ώστε να αποστείλουμε ένα απόλυτα σαφές μήνυμα και σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι δεν παίζουμε με το θέμα των βασικών δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι η υπηρεσία αυτή είναι μια εξωτερική υπηρεσία, ξέρουμε ότι θέλουμε να έχουμε μια ανθρωπιστική προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είμαστε σίγουροι ότι την χάνουν πλήρου σεβασμού ανά πάσα στιγμή. Ένα δεύτερο θέμα με το οποίο ασχολούν οι τροπολογίε είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία της Frontex. Ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να εισαγάγουν ε, αναφορές στις κατευθυντήριες γραμμές που ξέρουμε αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που σύνομα ελπίζω θα αποφανθεί πάνω στην ε, αξία των κατευθυνών γραμμών αυτών. Η δική μου πρόταση είναι ότι ενώ για την ουσία δεν έχω κανένα πρόβλημα να αφαιρθώ στην ουσία, στο περιεχόμενο των κατευθύνων γραμμών, τυπικά θεωρώ ότι δεν ήταν σωστό σε ένα νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισαγάγουμε μία αναφορά στο δικαστήριο που επιτίθεται, στο Συμβούλιο συγγνώμη, που επιτίθεται αυτή τη στιγμή μέσω του δικαστηρίου. Γιατί δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε μία απόφαση του Συμβουλίου που αυτή τη στιγμή ίσως θεωρηθεί μη ισχύουσα από το δικαστήριο. Έχουμε πάρα πολλές, ε, πολύ περισσότερες τροπολογίες ό,τι φανταζόμουν, αλλά για την προστασία των δεδομένων δεν είχαμε πάρα πολλές. Τούτο λεχθέντος είμαι ανοιχτό στο να προτείνω μια συμβαστική τροπολογία για το τμήμα που αφορά την προστασία των δεδομένων και που θα λαμβάνει υπόψη όσο δυνατόν περισσότερες ανησυχίες των συναδέλφων. Όσον αφορά την εκμίσθωση και την αγορά του υλικού. Η άποψή μου που συζήτησα και με τους Σκιώδης είναι ότι υπάρχει ευρεία συνένεση να ακολουθηθεί αυτή η άγουσα. Όσον αφορά τις επιστροφές και κατά πόσο θα μπορούμε να επιτρέψουμε στο Frontex να έχει και εκούσιες επιστροφέ και όχι, και και όχι μόνο εκούσιε, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί το θέμα. Τέλος, όσον αφορά το θέμα των τρίτων χωρών και συμφωνίε με τρίτες χώρες, υπάρχει νομίζω έντονη άποψη πολλών πολιτικών ομάδων ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής δημοκρατική, δημοκρατικός έλεγχος για το τι κάνει η υπηρεσία αυτή γενικά, αλλά ιδίως σε σχέση με τρίτες χώρες. Ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι προβληματικό για το Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά για να ξέρετε περίπου <clears throat> ε, ποιες, ποια είναι τα θέματα των απολογιών. Θα έχω και συναντήσει με τους κοιόδες με μονομένα ε, ομάδες και θα προσβλέπω τώρα στις απόψεις της Κομισιόν του Συμβουλίου και των συναντέλφων. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να κάνει ένα σύνομο σχόλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική εκθέση. Η εισήγησή του φαίνεται πολύ θετική και νομίζω ότι υπάρχει προοπτική να επέλθει συμφωνία. Αυτή είναι μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι είναι επίγουσα η κατάσταση ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τη Frontex άμεσα. Δεν μπορώ να αποφανθώ σε κάθε τροπολογία ξεχωριστά, αλλά θα σχολιάσω ορισμένα σημεία. Καταρχήν, νομίζω από πλευράς Κομισιόν ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη του ε, του εισηγητή σε σχέση με το ειδικό σώμα προστασίας ε, των συνόρων. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον επιχειρησιακό χαρακτήρα της πρότασης για να ενισχύσουμε την Frontex και να μην επιμείνουμε στο όνομα. Ο επιχειρησιακός χαρακτήρας έχει σημασία. Επ' αυτού θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν θα μπορέσουμε να δούμε τον ξεχωριστό κανονισμό ταχείας εφαρμογής που θα μπαίνει σε λεπτομέρειες, αλλά από όσο γνωρίζουμε από νομικής πλευράς ε, δεν ε, αποκλείεται να κινηθούμε προς την ε, κατεύθυνση που επιθυμεί ο εισηγητής. Ως προς τα προσωπικά δεδομένα έχετε την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για την στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας που θα βοηθήσει για οποιοδήποτε συμβιβασμό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ως προς ενδεχόμενες τροπολογίες. Α, δεν τελειώσατε, με συγχωρείτε. Επίσης, κατά την άποψή μας ως προς την εκούσια, τον εκούσιο επαναπατρισμό, όταν μιλάμε για συγκεκριμένα σχέδια ικανοτήτων των κρατών μελών, νομίζω ότι θα ήταν ε, επιθυμητό και θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο. Ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν προτεραιότητα για την Επιτροπή, δηλαδή να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα ως προς τη, τα, το νομικό πλαίσιο εφαρμογής. Θα επέλθει η πρόοδος νομίζω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Θα σταματήσω εδώ. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε και έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία ήδη από την πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ. Make a contribution. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ που μας δίνετε και την ευκαιρία να πούμε την άποψή μας για την ε, έκθεση. για τις ε, τροπολογίες που προτείνουν οι ευρωβουλευτές. Να πω καταρχάς ότι η έκθεση του κυρίου Μπουσούτηλ είναι πραγματικά εξαιρετική, μια εξαιρετική βάση, ε, μια εξαιρετική εκκίνηση για την πορεία. Και το συντομότερο δυνατό θα υποβάλουμε ένα σχέδιο συμβασμού. Ε, θα θέλαμε να γίνει αυτό κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Ε, πολλά από όσα ακούστηκαν από, τους, από τα μέλη της Επιτροπής σας δείχνουν την ε, βαθιά δέσμευση στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική, πιο ισχυρή Frontex. Συμφωνώ απόλυτα με, τον, με την πρόταση του κυρίου Μπουσούτιλ στην α, πρότασή του για την για το ότι θα πρέπει να γίνεται η, αναφορά στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα συγκεκριμένο άρθρο. Εδώ ο εισηγητής στην έκθεσή του κάνει αναφορά σε αυτό και εμείς το υποστηρίζουμε. Στην πρόσφατη συνάντηση της ε, ομάδας εργασίας για τη Frontex μιλήσαμε για κάποιες ε, ε που υπάρχουν ε. και εδώ πρέπει να πω ότι η πλειοψηφία των μελών ε, δέχονται ότι πρέπει να προχωρήσουμε ε, για τη Frontex και μάλιστα πολλοί έχουν ήδη ενσωματώσει τις ε, διατάξεις. Μετά την επόμενη συνεδρίαση σε, ομάδα, σε επίπεδο ομάδας εργασίας νομίζω ότι θα είναι έτοιμη μια πρόταση, ένα σχέδιο πρόταση εν πάση που θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τώρα, πάω στο θέμα της προστασίας των, δεδομένων. των δεδομένων. Θα γίνει και γι' αυτό μια πρόταση, ε, θα σας την υποβάλουμε. Μιλούμε για διάφορα εργαλεία και υποστηρίζουμε τα, το δημοκρατικό δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου προς τη Frontex και επίσης θέλουμε η συνεργασία της Frontex με τρίτες χώρες να διευρυνθεί. Προφανώς υπάρχουν και κάποιες εσωτερικές εκθέσεις οι οποίες βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου και είναι εμπιστευτικά έγγραφα, αλλά κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης που κάνατε χτες με τον Υπουργό, ε, είδαμε ότι η, ε, το να γίνουν αυτά τα, να πάψουν να είναι αυτά τα έγγραφα ε, εμπιστευτικά είναι λίγο δύσκολο ακόμη, αλλά η, η Προεδρία λέει ότι θα προσπαθήσει να είναι αυτά τα έγγραφα προσβάσιμα σε όλους, στα, σε όλα τα μέλη της, ομάδας, της Επιτροπής ΛΥΜΠ. Ε, επειδή έχουμε και άλλα μέλη που θέλουν να μιλήσουν, ε, ένα λεπτό ο καθένας και σας ζητώ να είστε σύντομοι γιατί μετά έχουμε και τους συντονιστές. Οπότε... Κάντε ό,τι μπορείτε. Για ένα λεπτάκι μόνο θα σα δίνω το λόγο, γιατί αλλιώ θα καθυστερήσουμε. Η κυρία Γκυγιόμ. Δύσκολο σε ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. Δεν θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε την εισηγήτρια της ΑΦΕΤ η οποία έχει ήδη εργαστεί στην ΑΦΕΤ πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αυτό προβλεπόταν και το νομίζω θα ήταν ε, ιδιαίτερα συνετό. Έχετε το λόγο. Thank you, uh, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχαμε ως κύριο μέλημα να δούμε πώς θα δομηθεί αυτή η γνωμοδότηση έτσι ώστε να βελτιωθεί η εργασία της Frontex για να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τώρα την πρόταση της Κομισιόν, η οποία κάνει την αναφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το θέτει ως προτεραιότητα, το οποίο επίσης ακούσαμε από την Κομισιόν, αλλά θεωρήσαμε ότι η πρόταση δεν ήταν, ε, ήταν πολύ περιορισμένη και δεν ήταν σαφής ως προς αυτό. Ε, έχουμε λοιπόν υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες και έχουμε συμφωνία στην ΑΦΕΤ για να υπάρξουν δεσμευτικοί και αποτελεσματικοί μηχανισμοί ώστε να γίνεται χρήση ανεξάρτητων και ποιοτικών, ανεξάρτητης και ποιοτικής εμπειρογνωμοσύνης ό,τι αφορά τα δεδομένα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και Όπω για παράδειγμα η υπατερμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε και για η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η αξιολόγηση της ε, υπηρεσίας, ε, η οποία δεν ήταν μέχρι στιγμής αναξάρτητη, και να συμπεριλάβουμε μία ανάλυση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία βασίζονται ε, στην χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστατεύονται. Και πρέπει να γίνεται ανάλυση, έχουμε πει, κάθε φορά που γίνεται αλλαγή, κάποια αλλαγή στον, στο καταστατικό της Frontex. δεν θα μπω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ένα θετικό είναι ότι οι Frontex και οι δραστηριότητες τους μπορούν να πάυσουν εάν σε περίπτωση που καταστατηγείται το ε, διεθνές δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε, ε, σας προτείνω να λάβετε υπόψη, να μελετήσετε όλες αυτές τις αλλαγές, γιατί είναι, γιατί είναι προτεραιότητα ενώ του Επιτρόπου να τροποποιήσει την, ε, την εντολή για τη Frontex για διάφορους λόγους. Ε, ένας από αυτούς είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις στην, ε, στα όσα γίνονται για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε είναι καλό που ακούμε ότι η Κομισιόν είναι ανοιχτή στην περαιτέρω συμπερίληψη τροπολογιών. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει μόνο μία παράγραφο να αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να είναι συγκεκριμένη και πρέπει να αναφέρεται. Σε όλα τα έγγραφα υπάρχει η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Ευχαριστώ. Εντάξει, τελειώσατε. Ναι, Madame Guillaume. Oui, merci. Κυρία Γκίγιομ, τι να κάνω, θα είμαι σύντομη κι εγώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουζούτιλ η διαδικασία με τους ε, σκιώδεις δεν έχει λήξει, θα επανέλθουμε επί ορισμένων θεμάτων. Θα ήθελα να υποστηρίξω τη σημασία αυτής της έκθεσης που απαιτέλεσε αντικείμενο σωρίας τροπολογιών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα αναφερθώ σε ορισμένες ως προς τα βασικά σημεία δηλαδή. Ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι ζωτική σημασίας, ε, εφήγησαν ερωτήματα από πολλούς και σχηματικά είπαμε κατά πώς θα πρέπει να υπάρξει μία ειδική παράγραφος με πολλές ε, μνήες. Νομίζω ότι πράγματι θα πρέπει να προβλέψουμε μία αρχική παράγραφο αρκετά εκτενή που να αναφέρεται στα θεμολιώδη δικαιώματα για να αποστέλουμε ένα μήνυμα ως προς το περιεχόμενο αυτό του κειμένου, ότι προσδίδουμε δηλαδή μεγάλη σημασία στα θεμελιώδη δικαιώματα και μετά να υπάρχουν μία κλειδιά. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που θα πρέπει να μνημονευθούν ιδιαίτερα ως προς την κατάρτιση της επιχειρήσης και όταν μιλάμε για αξιωματούχους συνδέσμους θα πρέπει να ε, μιλάμε, να δίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τη σύνθεση αυτού του σώματος. Κύριε Λόχ Μπίλερ μας έδωσε σωστές κατευθυντήριες γραμμές. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσα στα πλαίσια νομικής διαφάνειας για να θέσουμε σε εφαρμογή άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μιλώντας για τη Frontex, για τα προσωπικά δεδομένα, ο κύριος ε, Μπουζούδηλ προσδίδει ε, σημασία σε αυτό το θέμα, αλλά εν περιπτώσει η εντολή της Frontex αφορά την εξέταση των προσωπικών δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω όμως ε, γιατί πρέπει να χρησιμοποιεί ευρέως τα προσωπικά δεδομένα. Μιλάμε για καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς την χρήση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει ένα στενό πλαίσιο ε, ερμηνείας. Ως προς τη δημοκρατική εποπτεία έχει επιτελεστεί πρόοδος και στο ποσοτικό, ως προς το ποσοτικό και το ποιοτικό σκέλος, ιδιαίτερα ως προς τον εκούσιο επαναπατρισμό. Η Frontex έχει μια εντολή για τον εκούσιο επαναπατρισμό και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ανάκτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων που αναλαμβάνει η Frontex. Ως προς την αγορά ή το leasing, εδώ αντιτάσσουμε τον δαπανηρό χαρακτήρα το, του εγχείρηματος αυτού και δεν θέλω να φανεί ότι κατασπαταλούμε χρήμα. Θέλουμε να αυτονομήσουμε κάπως ε, τη Frontex μέσω αυτής της έκθεσης, το κατανοούμε αυτό, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ορισμένες διευκρινήσεις ως προς τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες της Frontex. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια συμφωνία επί του θέματος. Bene. Signora Thank you very much. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσούτιλ για την ε, πραγματικά πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Ακέραιη και ε, ε, αξιέπαινη και συγχαρητήρια και στους συναδέλφους που ήταν οι σκιώδες Και εγώ θα ήθελα να τονίσω την ε, σημασία μιας στενής συνεργασίας ε, εδώ στο Νίκο μας για να έχουμε τελικά μια, ένα σωστό δομημένο κείμενο, να είναι σαφή τα επιχειρηματά του που θα πάει στο Συμβούλιο και στην ίδια τη Frontex. Πολλές από τις τροπολογίες, έχουν που, που χρειάζονται να τις μελετήσουμε και είναι σημαντικό να μην βιαστούμε. Είναι σημαντικό οι αποφάσεις, με, να, μας να έχουν μία στέρεα βάση και να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε συμβιβασμούς στους οποίους να μπορούν να υποστηρίξουν όλες οι ομάδες έτσι ώστε το κείμενο μας να έχει την απαραίτητη βαρύτητα. Έχουν υπάρξει πολλά σημαντικά στοιχεία τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι. Εγώ θα περιοριστώ να πω τα εξή. Η πρόταση, ας πούμε, του κυρίου Μπουσούτιλ να βάλουμε μια ταμπέλα, μια ετικέτα στο ε, σύστημα, στο, ε, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι λίγο θέμα διατύπωσης. Ε, η ιδέα που κρύβεται από πίσω νομίζω είναι αυτή ακριβώς που λέει ποιες είναι οι δραστηριότητες της Frontex και νομίζω ότι θα είναι δεκτική από τη Frontex. Εγώ θα την υποστηρίξω. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να διαφωνούμε τώρα για, τέσα, για τόσα μικρά πράγματα. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά προστασία δεδομένων, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Τώρα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες της Frontex πάντα θα σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μα γι' αυτό ακριβώς μπήκε αυτή η μεγάλη τροπολογία σε αυτή την έκθεση. Θα μπορούσε ίσως και να διευρυνθεί. Νομίζω γίνεται αυτό. Αλλά πρέπει να τονίζουμε ότι όλοι οι συνοριαφύλακες που δουλεύουν στη Frontex πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Επίσης χρειάζονται και ε, συγκεκριμένη εκπαίδευση ως προς αυτό. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να δώσουν την ε, καλύτερη ε, υποδοχή στους, ε, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, ειδικά όταν βλέπουμε ότι κάποιος έχει ανάγκη η ετάτε ασύλου. Αυτό πρέπει να είναι πάντα και το ότι θα πρέπει να γίνονται αυτά τα δικαιώματα του βέβαια πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό μας. Αυτό είναι το, το πρώτο και το βασικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Καλωσορίζω την ε, γνωμοδότηση της, της ΑΦΕΤ που ψηφίστηκε πρόσφατα και χαίρομαι που άλλαξε ο όρος ε, illegal migrants και έγινε irregular migrants. Και άλλοι ε, συναδελφοί έχουν ε, το έχουν προτείνει αυτό. Ελπίζω και εδώ στη Λίβη να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Ε, τα, μπορεί, οι άνθρωποι σίγουρα ποτέ δεν είναι παράνομοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα αγαστής συνεργασίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή ότι υπάρχουν 7 ομιλητές. Δεν πρέπει να ξεπεράσετε το 1,5 λεπτό κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσούτιλ. Σπάνια κάνουμε τόσο καλές συναντήσεις ισκιώδης, με τόσο καλή δομή, με τόσο καλές συζητήσεις και το ότι μπορούμε να συζητάμε όλα αυτά και να, τα, να φέρνουμε τόσο καλά αποτελέσματα στην Επιτροπή είναι εξαιρετικό. Πολλά συγχαρητήρια. Οι άποψεις μου δεν διαφέρουν από αυτές των συναδέλφων. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μία κοινή δήλωση για τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την τήρησή του, το σεβασμό του και το πρόβλημα που υπάρχει στον τομέα αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε και στις αιτιολογικές σκέψεις να πούμε ότι θα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο άρθρο ως προς αυτό. Και επίσης θα πρέπει να δούμε και στο διατακτικό σε ποιο σημείο είναι απαραίτητο, είναι υποχρεωτικό να έχουμε συγκεκριμένες διατυπώσεις για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό εντάξει μπορούμε να το δούμε, δεν είναι τρομερό. Ε, αυτό είναι το πρώτο. Ένα δεύτερο σημείο ε, για την εθελούσια επαναπατρισμό. Ε, το ξανασκέφτηκα και εγώ, είδα και στην δική μου ομάδα τι γίνεται. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ε, ας μην αναμειγνύουμε τα πράγματα και αν δούμε και την ε, ε, ε, εντολή της Frontex δεν νομίζω ότι ταιριάζει κάτι τέτοιο εδώ. δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το πρόβλημά μου, και το είχα πει στη συνάντηση, ο όρος Frontex, ε, ομάδα υποστήριξης, ε, έτσι ε, προέκυψε ξαφνικά, είμαστε σε ένα, έχουμε τώρα ένα σύστημα προστασίας συνόρων, είναι λίγο δύσκολο γιατί ούτως ή άλλως εμείς έχουμε πρόβλημα με την Frontex, νομίζω λοιπόν δεν μπορώ να το, να το δεχτώ αυτό. Και μια τελευταία σκέψη για τους τεχνικούς εξοπλισμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών. Γιατί υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα ακόμη εκκρεμή, τα οποία όμως τώρα δεν θα ήθελα να θέξω. Ευχαριστώ. Σένα Φλότρο. Φλότρο. Ευχαριστώ. Για να αναφερθώ στα σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο Σιμών Ζούτιλ μίλησε για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, είναι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της αναθεώρησης του κανονισμού Frontex. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν γενικές ρήτρε σε όλα τα άρθρα σύμφωνοι, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε και επιχειρησιακούς μηχανισμούς έμπρακτα έτσι ώστε οι ρήτρες για την διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορούν να εφαρμοστούν έμπρακτα. Υπάρχει μία ε, έξοχη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη σχέση μας με την Τινησία, όπου είχαμε ένα, μια κυβέρνηση διαφθοράς που λειτουργήσε εξαιρετικά πάνω από 10 χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι να εγγυηθούμε την ύπαρξη ορισμένων μηχανισμών έτσι ώστε η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ε, προλαμβάνεται ή εν πάση περιπτώσει όταν διαπιστώνεται να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ είναι θέμα ευθύνης διότι εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση νοχέλιας για το τι μπορούμε να αναθέσουμε στα κράτη-μέλη ή στη Frontex σε περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δική μου ομάδα ε, υποβάλλει μία πρόταση που θα ήθελα να εξετάσετε. που αφορά τα άρθρα 245 και 246 μετά από διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναθέσουμε ή να αποδώσουμε ευθύνες στα πλαίσια διασφάλισης ενός συμβολέου με μια τρίτη χώρα ή εάν δεν υπάρχει συμβατικός χαρακτήρας μιας επιχείρησης της Frontex. Δηλαδή, να αποσαφηνίσουμε μια κατάσταση για να μην παραμένει συγκεχημένη. Δηλαδή να αυξήσουμε αρμοδιότητες, αλλά θα πρέπει να διασαφηνίσουμε θέματα απόδοσης ευθυνών. Ως προς το μηχανισμό αυτό υπάρχουν θέματα κατάρτισης, ανάλυσης κινδύνου, επιχειρησιακών σχεδίων, μιλάμε για κατάρτιση πρωτίστως, για κώδικα συμπεριφοράς, έτσι ώστε να αποφύγουμε ανθρώπινα δράματα. Επίσης, εάν δεν υπάρχει ε, αυτόνομη παρατήρηση, δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις συμβατικές και μη ευθύνε ως προς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ετούντες άσυλο. Θα ήθελα ο εισηγητής να λάβει υπόψη όχι μόνο ωραία λόγια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μηχανισμούς Κολέγια Κολέγα Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ πολύ, με πολύ προσοχή τη συζήτηση που κάνουμε και έχω διαβάσει με πάρα πολύ προσοχή όλες τις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε ότι κατάγομαι από την Ελλάδα, μια χώρα που δέχεται αυτή την περίοδο τη μεγαλύτερη πίεση σε σύγκριση με ε, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και θέλω στο σύντομο χρόνο που έχω να ε, κάνω ορισμένε πολύ σύντομε παρατηρήσεις. Το πρώτο, ε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μπουζουτήλ για την εξαιρετική του έκθεση, μια έκθεση η οποία καταρχήν αποτελεί μια πολύ αξιόπιστη βάση για να μπορέσει η Frontex να ενισχυθεί, να έχει καλά αποτελέσματα και βεβαίως να διασφαλίσουμε και όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα και νομίζω ότι ε, και με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες έχει, έχει συνεργαστεί εξαιρετικά. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σας μεταδώσω τι συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή την περίοδο στο ε, πολύ λίγο χρόνο που έχω. Ξέρετε, αν ρωτήσετε έναν Έλληνα σήμερα ποια είναι η μεγαλύτερη συνδρομή της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ιδίω αυτή την περίοδο, επειδή ξέρετε πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι νιώθουν καταλελειμμένοι σε σχέση με την αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε, η απάντηση που θα πάρετε από τους περισσότερους σε ό,τι αφορά την πραγματική αλληλεγγύη της Ευρώπης είναι η Frontex η Frontex ήρθε στον Πειραιά, είναι στο Αιγαίο και κάνει επιχειρήσεις. Ήρθε τώρα και με τα Rabbits στα ε, σύνορα τα χερσαία με την Τουρκία και, ε, και παρουσιάζει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και βεβαίως πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Και θέλω να πω, ακριβώς επειδή στην Ελλάδα παρακολουθούμε όλη τη Frontex, και επαναλαμβάνω ότι σέβομαι απολύτω όλα τα επιχειρήματα που έχουν τεθεί και ελπίζω να καταλήξουμε ε, σε ένα, κοινό τόπο και να συμφωνήσουμε όλοι δεν έχουμε ακούσει κάποια καταγγελία για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων το λέω σε ό,τι αφορά τη δράση τη Frontex στη δική μου χώρα καμία, καμία καταγγελία Αντιθέτω, οι αναφορέ που γίνονται είναι σε ό,τι αφορά την επικοδομητική συνδρομή τη Frontex και στι επιχειρήσει αλλά και στην ε, μεταφορά τη τεχνογνωσία. Ε, Αυτά θέλω να πω καταρχήν και να παρακαλέσω συμπερασματικά αυτό κύριε Πρόεδρε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αφού συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη Frontex, να συνεχίσουμε να την καθιστούμε εξίσου αποτελεσματική και ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που και όλες οι άλλες πολιτικές ομάδες ήταν τόσο ικανοποιημένες με τον Σάιμον Μπουζουτήλ. Και εμείς το ίδιο. Και θα ήθελα να τον καλέσω πραγματικά να σας καλέσω όλους να υιοθετήσετε αυτά που λέει και από τις ουσίες γιατί είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, εδώ συζητάμε τώρα την ενδυνάμωση του Frontex. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει και γι' αυτό θα πρέπει να επεξεργάζεται τα στοιχεία, βέβαια υπό την προστασία των δεδομένων και του κανόνε που υπάρχουν σχετικά και λαμβάνοντα υπόψη τα βασικά δικαιώματα. Νομίζω ότι μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να βοηθήσουμε ούτως ώστε η Frontex στην αξιολόγηση και επιτήρηση ίσως ε, του κεκτημένου Σέγγεν να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά το κείμενο της Κομισιόν, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πολύ εξαρτάται ακόμα το Frontex από την έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχει δύο ε, ψήφους στη Διαχειριστική Επιτροπή για να μπορέσει έτσι να επιδράσει και αυτό εξασφαλίζεται και από τον θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ευηρεξία στη Frontex, κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κύριε Κέλλερ. Ευχαριστώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δραστηριότητε του Frontex στην ε, Ελλάδα. Έχουμε ορισμένες εκεί που ήταν ότι πραγματικά ε, στη Γερμανία, Γερμανούς δηλαδή που είναι στα σύνορα εκεί και που είδαν πόσο απέσες είναι οι προϋποθέσεις διαβίωσης των μεταναστών. Για τις δραστηριότητες του Φρόνταξ, λέω. Ναι, ναι, αυτό λέμε. Έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Οπότε κατάλαβα μια στιγμή, η Κομισιόν δεν ε, έχει πολλές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων στην πρόταση γιατί είπε η Κομισιόν ότι εμείς δεν θέλουμε να προβλέψουμε να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα οι υπηρεσίες Frontex. Τώρα είπατε ότι θέλετε μία βελτίωση, ε, είπατε ότι ο κ. Μπουσουτήλη θέλει επίσης να προβλέψει, δηλαδή εσείς θέλετε η Frontex να επεξεργάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τι εννοείται με αυτό. Κοράτσα Μπίλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να σας υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τις θαλάσσιες ε, επιχειρήσεις που συντονίζει η Frontex όταν ελήφθη η απόφαση του ε, Συμβουλίου υπήρχε συμφωνία σε όλες τις πολιτικές ομάδες για την ανάγκη για σαφείς κανόνες για να εξετε... αντιμετωπίσουν επίγουσε καταστάσεις ενδεχομένω στη θάλασσα. Για τους λόγους που μας υπενθύμησε ο Σάιμον, γιατί υπάρχει μια εκδημούσα υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και κατά πόσο αυτό θα το εδώ στο κανονισμό, ναι, έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία και θα ήθελα να παρακαλέσω του αδέρφου να την υποστηρίξουν, δηλαδή τροπολογία παριθμών 70 θα πρέπει να προβλέψουμε να γίνονται σεβαστές οι εκκρεμούσες διαδικασίες και θα ήθελα να ε, συμφωνήσετε μαζί μου επί της ουσίας να έχουμε σαφείς κανόνες. Και εγώ εντάχει θα ήθελα να πω μερικά λόγια ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του Σάιμον Μπουζούτιλ γιατί πραγματικά ε, έμπρακτα πρόθυσε όλα τα ζητήματα που αφορούσαν όλες τις πολιτικές ομάδες. Και αυτό ισχύει και για τις ε, τροπολογίες. Μιλάμε για έναν οργανισμό τον οποίο θα πρέπει να ελέγχουμε, να δούμε ποιες είναι οι δαπάνες και ποια είναι η απόδοση. Τώρα αλλάζουμε τον κανονισμό γιατί οι μηχανισμοί αντιστάθμισης δεν ε, λειτουργήσαν καλώς. Μιλώ για τη συνεργασία με τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και τον Frontex. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ταχείας επέμβασης, επέμβασης στα σύνορα και να υπάρχει και η ε, δυνατότητα κατάσχεσης. Εάν μιλάμε για πραγματικά παραπτώματα, θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κατασχεθέντα τα οποία να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια σε ενδεχόμενες προσφυγές. Και επίσης έχει σημασία να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Πριν δώσω το λόγο στο Σάιμον Μπουζούτιλ, θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή μετά από το ερώτημα που έθεσε η συνάδελφος Κέλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η Κομισό δεν άλλαξε άποψη. Θα πρέπει να είναι σαφή τα πράγματα. Στην αρχή, όταν υιοθετήσαμε την πρόταση, είχαμε κατά νου να εξετάσουμε το θέμα των προσωπικών δεδομένων και η Κομισιόν τότε αποφάσισε να εξετάσει το θέμα εις βάθος. Και γι' αυτό, αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν είχε αναφέρει το θέμα των προσωπικών δεδομένων στην αρχική της πρόταση η Κομισιόν. Αλλά όπως είπε όταν υιοθετήθηκε η, η πρόταση της Κομισιόν για το κανονισμό Frontex, είπε ξεκάθαρα λέει η Κομισιόν τότε ότι το εξέταζε το θέμα και ότι αν χρειαζόταν θα πανέρχετο και θα συνέβαλε στην ε, συζήτηση με όλα τα στοιχεία για όλα τα συστήματα ενημέρωσης που υπήρχαν. Και μόνο μετά από αυτό <clears throat> μπόρεσαν να καθοριστεί η συμμετοχή στη συζήτηση και ο τρόπος με τον οποίο προχωράνε τα πράγματα. Εάν χρειάζεται θα έχουμε επικοδομητική συζήτηση. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανένα ότι άλλαξε άποψη η Κομισιόν για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σάμον Πουζουτήλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα συγχαρητήρια και τα εγκόμια τους. Εάν θα ήθελα να κρίνω το αποτέλεσμα πάνω στο φάκελο αυτό βάσει των συγχατηρίων θα είχαμε οπωσδήποτε ομοφωνία στην Επιτροπή. Αλλά καταλαβαίνω τα πράγματα είναι κάπω πιο πολύπλοκα. Και γι' αυτό θα χρειαστούν πολλέ περισσότερε συζητήσει. Θα ήθελα να αναφερθώ σε λίγα συγκεκριμένα θέματα. Ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αυτό το σημείο της κυρίας ε, Φλότρο, ότι χρειαζόμαστε έναν λειτουργικό μηχανισμό για να είμαστε σίγουροι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ελέγχονται επαρκώς. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο μου άρεσαν οι τροπολογίες των φιλελευθέρων που ακριβώς προτείνουν τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής που θα συμπεριλαμβάνει και άλλους ε, ε, εκτός του Frontex. Είμαι ανοιχτό όμω, να λάβω υπόψη και άλλα στοιχεία και να λάβω υπόψη την παρατήρηση της κυρίας Λόχ Μπίλερ να σταματήσουν δηλαδή οι επιχειρήσεις εάν υπάρχουν αποδεδειγμένες παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να περάσω σε κάτι που είπε η κυρία Γιγιόμ. Είναι αληθές ότι εκ πρώτης όψης μπορεί κανένας να αναρωτηθεί γιατί μια υπηρεσία όπως η Frontex θα πρέπει να επεξεργαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά είχατε έρθει στη Βαρσοβία και ξέρουμε ότι διευκρίνησε απόλυτα η υπηρεσία αυτή ότι παρόλους τους πόρους και τα μέσα που τις διαθέτουμε καμιά φορά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που οι συλλέγεται σε αποστολέ για τι οποίε όλοι, όλοι πληρώνουμε. Και επειδή δεν μπορεί να επεξεργαστεί τι πληροφορίε αυτές, δεν μπορεί να ε, ασκήσει το, να πραγματοποιήσει μάλλον το έργο της μέχρι τέλους. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτή γιατί δεν έχει την, την νομική βάση. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και αυτή τη δυνατότητα εφόσον ε, συμμετέχει η EDPS. Αυτό δεν με προβληματίζω. Ελπίζω λοιπόν ότι για την προστασία των δεδομένων θα μπορέσουμε να πτύχουμε συνένεση. Τουλάχιστον μεγάλη πλειοψηφία. Αυτά. Ελπίζω και θα συνεχίσω να εργάζομαι ούτω ώστε να επιτευχθεί κατά τη δυνατόν ευρεία υποστήριξη του φακελού και μόνο γιατί όπως είπε η Συρία Βίξερο, ότι αυτό θα ενδυναμώσει το Κοινοβούλιο στην αντιμετώπιση του, του Συμβουλίου. Ας μην είμαστε απλοϊκοί αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι το Συμβούλιο θα είναι πιο μινιμαλιστικό στις απαιτήσει του για το φάκελο αυτό. Λοιπόν, όσο πιο ισχυρή είναι η πλειοψηφία, τόσο πιο ισχυρή θα είμαστε στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο ελπίζουμε, α φτάσουμε σε μια συμφωνία πρώτη ανάγκη, Όπω είπε ο Γιώργο χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό Frontex. Όχι αύριο. Ούτε καν σήμερα. Χθε. Χθε. Κάτι πηγόντω. Τέλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και ιδίω την κυρία που είναι δίπλα σα, κύριε Πρόεδρε, γιατί χωρί την υποστήριξη τη Γραμματεία, πολλό από το έργο που επιτελούμε δεν θα ήταν δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, βεβαίως και ως προς το τελευταίο που αναφέρατε όλοι συμφωνούμε. Μετά από την ζωηρή συζήτηση και άκρος ενδιαφέρουσα θεωρούμε ότι κατά τα μέσα Μαρτίου θα ψηφίσουμε γενικά για αυτό το θέμα και στο μεταξύ ο κύριος Μπουζούτιλ θα έχει επαρκή χρόνο για να μπορέσει να ορίσει με τους σκιώδεις, να επεξεργαστεί μάλλον τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού. Θα έπρεπε να συζητηθεί κι άλλο ένα σημείο, αλλά έχουμε ξεπεράσει την ε, ώρα μας, το ωράριο εργασίας, γι' αυτό κλείνει η συνεδρίαση και τώρα θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Καλό μεσημέρι.